Καλησπέρα σας. Σε όλες τις γλώσσες καλησπέριζει ο Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θα ήθελα να να καλωσορίσω σε αυτή την κοινή συνεδρίαση Επιτροπής Απασχόλησης και Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών τους πάντες και πριν ξεκινήσουμε με την πρώτη ψηφοφορία στο πρόγραμμά μας θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται μέχρι το πέρας της συνεδρίασης. Δεύτερον, I would like you to endorse the coordinator's recommendation. Θα ήθελα να εγκρίνουμε και την σύσταση των συντονιστών για τους ε, εισηγητές, για τις εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις που συμφωνήσαμε στις συνεδρίες των συντονιστών. Έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης είναι για την κυρία Γκυγιόν. Εισηγήτρια κυρία Γκυγιόν γνωμοδότηση για τη Συμφωνία ε, Παραποιημένων Προϊόντων Εμπορίου, ε, συντάκτης ο κύριος Δρούτσας, έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθαρίζει ως τμήμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ε, το μέσο για τη χρηματοοικονομική στήριξη για τα εσωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις. Το αναλαμβάνει ο κύριος Μαρινέσκου πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο τμήμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ένα μέσο για τη χρηματοοικονομική στήριξη για την καταπολέμηση του εγκλήματος ε, και τη συνδρομή στις αστυνομικές δυνάμεις. Ο κύριος Ιακολίνο αναλαμβάνει τη σχετική έκθεση. Και τέλος, προστασία κρίσιμων πληροφοριών και υποδομών. Η κυρία Χάνκη. Εάν συμφωνείτε λοιπόν, μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε με την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα καταρχάς να πω σε όλους σας, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ότι όπως συμφωνήσαμε στις συνεδρίες των συντονιστών, Θα θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στον κύριο Εμίλιο Ντικαπιτάνη για την μακρά του καριέρα και πορεία, ο οποίος ε, υπηρέτησε την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για πάνω από 20 χρόνια και συνταξιοδοτείται λόγω ηλικία και συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής για τα όσα κατάφερε με σύνεση, σοφροσύνη και ε, για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάντα διατεθειμένος να συνεργαστεί μαζί μας ανεξάρτητα από το πολιτικό κόμμα και την πολιτική οικογένεια στην οποία ανήκε. Για άλλη μια φορά λοιπόν, του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τον βλέπουμε και στο μέλλον και βεβαίως Ελπίζουμε ότι αυτός που θα τον διαδεχθεί ως επικεφαλής του Τμήματος ε, Νομικών Θεμάτων για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα έχει τα ανάλογα προσόντα. We are now... Και τώρα να σας πω ότι η ψηφοφορία για την γνωμοδότηση Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Υπηκότητα για την άρση των προσκομμάτων για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών έχει αναβληθεί σε συμφωνία με την εισηγήτριά μας, την κυρία Ντάνοκα και ναι, μεν δεν θα γίνει συγκεκριμένη ψηφοφορία, αλλά έχουμε άλλες τρεις. Η ψηφοφορία που αναβλήθηκε θα γίνει εν ευθέτω χρόνο, θα σας ανακοινωθεί η ημερομηνία. Να σας υπενθυμίσω ότι θα κάνουμε και ηλεκτρονική ψηφοφορία, γι' αυτό ε, βεβαιωθείτε ότι έχετε την ηλεκτρονική σας κάρτα. Όποιος δεν έχει την κάρτα του, σας παρακαλώ να στείλει κάποιον να τη φέρει, διότι ψηφίζουμε. The first vote. Πρώτη ψηφοφορία στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Πολιτικών Ελευθεριών και Απασχόλησης βάσει του άρθρου 50 του κανονισμού του Κοινοβουλίου είναι η διαδικασία ενιαίας αίτησης για άδεια παραμονής και εργασίας. Η συγγήτρια για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών είναι η κυρία Βερονίκ Ματιέ και η Συνδεδεμένη Επιτροπή έχει τον Αλεχάνδρο Σέρκας ως ε, συνεισηγητή. Θα ψηφίσουμε λοιπόν για την έγκριση της συμφωνίας αυτής και τις τροπολογίες για τη δεύτερη ανάγνωση. Στη δεύτερη ανάγνωση θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία και η κυρία Λίν είναι εδώ ως συμπεριοδρεύουσα για την ε, ψηφοφορία αυτή. Δεν ξέρω αν θέλετε το λόγο από πλευράς Επιτροπής Απασχόλησης. Όχι. Ιδάλλως λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία αυτή. Yes. It's, it's an orientation vote. Πρόκειται για ψήφο προσανατολισμού. Γι' αυτό λοιπόν Δεν χρειαζόμαστε ηλεκτρονική κάρτα. Ψήφος προσανατολισμού. Υπέρ. Those against. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν θετική ψήφος. Ζητά έλεγχο μία συνάδελφος, επομένως μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το πρόβλημα the problem Υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης που συμμετέχουν στη σημερινή συνεδρίαση πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ως ε, μέλη που ψηφίζουν για αυτή την κοινή ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Ωραία. ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Now the vote is closed. Πέρασε της ψηφοφορίας. We have here 40 plus. 40 υπέρ, 3 κατά, 23 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν ο ψήφος προσανατολισμού. Προχωρούμε. Only leaving. Only leaving. Now We're going to have a second vote on this. Και τώρα θα ψηφίσουμε για δεύτερη φορά στο θέμα αυτό, αλλά μόνο για τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Μόνο λοιπόν για τα μέλη της ΛΥΜΠΕ. It seems that the electronic system is not ready yet. Φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμο ακόμα το ηλεκτρονικό σύστημα. Περιμένουμε λιγάκι και θα συνεχίσουμε. Not yet. Μόνο τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ψηφίζει για το σχέδιο σύστασης για δεύτερη ανάγνωση. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε της ψηφοφορίας. Among the members, 29 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, 12 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Shall we go now for the second thing?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 λίγο την προσοχή σας. Η Επιτροπή Απασχόλησης αποχωρεί από την αίθουσα και καλώ τους υπολείπους να παραμείνουν γιατί έχουμε μια δεύτερη ψηφοφορία. Περνάμε τώρα σε μια ψήφο για, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Και πάλι βέβαια θα πρέπει να συγχαρούμε τις δύο συνεισηγήτριες και τους κοιόδης εισηγητές διότι συνεισέφεραν ιδιαίτερα στην προστασία των θυμάτων και ευχαριστούμε και την Επιτροπή Γυναικών για τη συνεργασία βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και τον κύριο Γκούσταυσον, ε, πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών ε, και Ίσων Δικαιωμάτων. Αν θέλετε να πείτε δύο λόγια, Παρακαλώ, αλλιώς θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ξεκινά λοιπόν η ψηφοφορία. Ψήφος προσανατολισμού. Μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέραση ψηφοφορίας. 46 plus. 46 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, Καμία αποχή. Συγχαρητήρια λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι. Συγχαρητήρια στις συνεισηγήτριες και στους κοιόδης εισηγητές, ευχαριστούμε και τον κύριο Γκούσταυσον. Και έχουμε και μια τρίτη ψηφοφορία. We are still a third vote here. Υπάρχει τρίτη ψηφοφορία, σας παρακαλώ. Let's do it the sooner the better. Now we're Ψηφίζουμε τώρα λοιπόν το σχέδιο έκθεσης. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροποποίηση του κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό που θεσπίζει ένα κοινοτικό κώδικα θεωρήσεων. Η συγητής είναι ο κύριος Λουί Μισελ. Σας ευχαριστούμε πολύ για το έργο σας. Και προχωρούμε με την ψηφοφορία. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Περιμένουμε μισό λεπτό για να ξαναξεκινήσει το σύστημα. We are waiting for a second. Nope. Okay, now we got the signal. The vote is open. Λοιπόν, ε, έχουμε σήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη, μισό λεπτό να ανακοινώσω τις τροπολογίες. Τροπολογία υπεριθμών 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη 11 τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Και τώρα το κείμενο ως τροποποιήθηκε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε της ψηφοφορίας. 39 ψήφοι υπέρ. Δύο ψήφοι κατά, μηδέν εποχές. Ευχαριστούμε κύριε Μισελ, σας συγχαίρουμε. Σας ευχαριστώ όλους. And now, having come to an end, Επειδή λοιπόν ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης, ο απολογισμός της Πολωνικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Περιμένουμε λοιπόν τους Πολωνούς υπουργού. Παρακαλώ. Monsieur Michel, à la prochaine. Hi.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 Προχωράμε παρακαλώ. work. Συνεχίζουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Καταρχάς να καλωσορίσουμε τον κύριο Ίγκορ Τζιάλουκ. Ελπίζω να πρόφερα το όνομά σας σωστά. Παλιός φίλος και υφυπουργός ε, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μαζί του θα είναι ο κύριος Πιότρ Στασάνσκικ, Σταχάνσκικ, υφυπουργός του Υπουργείου Ιστορικών. Εκπροσωπούν την Πολωνική Προεδρία του Συμβουλίου και είναι εδώ σήμερα για να παρουσιάσουν τα συμπεράσματα της Πολωνικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης ε, και στη συνέχεια θα έχουμε ε, μια διαδικασία ερωταποκρίσεων. Στη συνέχεια θα έχουμε, αφού ακούσουμε τον κύριο Τζιάλου, τον κύριο Σταχάνσκι, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Πολωνικής Προεδρίας στον τομέα της ασφάλειας και των ιστορικών υποθέσεων. Ε, και πάλι θα υπάρχει γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων. Κύριε Τζιαλούκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τα καλά νέα είναι ότι τελειώνει η Πολωνική Προεδρία και θα μας ε, ξεφορτωθείτε με αυτά τα δύσκολα, τα ονόματα που δεν μπορείτε καν να προφέρετε. Ελπίζω βέβαια να έχετε και κάποιες καλές αναμνήσεις από την Προεδρία μας. Εξαιρετικές. Μπορείτε να βάλετε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω τη μητρική μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, την Επιτροπή ε, για την ε, σημερινή πρόσκληση είναι τιμή μου. Θα εκπροσωπήσω την Πολωνική Προεδρία και θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ε, ότι τους τελευταίους έξι μήνες είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ήταν η πρώτη Πολωνική Προεδρία και άρα μια πολύ σημαντική πρόκληση για μας υπήρχαν υψηλότατες προσδοκίες από πλευράς των πολιτών της Ένωσης από όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ' τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας στήριξε σε μεγάλο βαθμό στις εργασίες μας. Επανειλημμένα η Επιτροπή εξέφρασε την υποστήριξή της για το έργο της Πολωνικής Προεδρίας και αυτό επιβεβαιώνεται από την έκβαση της σημερινή ψηφοφορία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασία. Είναι ένα μόνο παράδειγμα τη αγαστής συνεργασίας που είχαμε με το Κοινοβούριο και συγκεκριμένα με την Επιτροπή σα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητέ ε, για την έκθεση αυτή. Κατά τη διάρκεια της ε, Πολωνικής Προεδρίας θελήσαμε να αλλάξουμε την προσέγγιση που υιοθετούμε ως προς το ποινικό δίκαιο. Μέχρι τούδε εστιάσαμε την προσοχή μας ε, στα κατασταλτικά μέτρα. Κατά των ε, δραστών των αξιοπίνων πράξεων. τώρα, θα θέλαμε να ασχοληθούμε και στη, τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας με τα δικαιώματα των θυμάτων. Είναι ύψιστη προτεραιότητα για μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και μπορώ να σας πω σήμερα ότι ήδη έχουμε σημειώσει επιτυχίες και χαίρομαι που υποστηρίξατε τη θέση και το έργο μας επειδή αναγνωρίσατε την αναγκαιότητα αυτής μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας για μεγάλο αριθμό φακέλων και για άλλους έχουμε ρίξει τα θεμέλια για τις επόμενες προεδρίες. Ορισμένα θέματα εκκρεμούν. Ευελπιστούμε το επόμενο δεκαήμερο ε, και συγκεκριμένα στην, ε, στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης θα μπορέσουμε να κλείσουμε και άλλους φακέλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την αίσια έκβαση της ε, ψηφοφορίας σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Όπως και η Ισπανία, έτσι και η Πολωνία ανέκαθεν υποστήριζε την προσπάθεια αυτή και πιστεύουμε πραγματικά ότι τα θύματα θα τύχουν καλύτερης προστασίας χάρη σε αυτό το σχέδιο οδηγίας. Θα προστατευτούν καλύτερα κατά της καταχρηστικής συμπεριφοράς. Θα προστατευτούν από τους αυτοργούς των εξέπινων πράξεων. Ξέρουμε ότι οι εγκληματίες δεν πρόκειται να τους κυνηγήσουν σε άλλε χώρε της Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα θύματα γνωρίζουν ότι θα έχουν μια επαρκή προστασία η Κάρμεν Ρομπέρο Λόπες και η Τερέσα Χιμένες Μπεθερίλ εργάστηκαν σκληρά και χωρίς τη δική τους ε, συμμετοχή. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Θα ήταν ε, πολύ πιο χρονοβόρη η διαδικασία έγκρισης του σχεδίου οδηγίας. Καταφέραμε να υπερπηδήσουμε τα προσκόμματα τα κολλήματα που είχαν δημιουργηθεί, ε, που προέκυπταν αν θέλετε και από τη συνθήκη. Και μετά από ε, δύο χρόνια δουλειάς και για το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουμε πλέον προγραμματίσει την υπογραφή για έχει προγραμματιστεί η υπογραφή για την 3η ε, Δεκεμβρίου, πρώτη συνόδου κορυφή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων θα ήθελα να απευθύνω μία έκκληση προς την ε, ε, επόμενη Προεδρία ε, να συνεχίσει τις προσπάθειές μας στα θέματα αστικού και ποινικού δικαίου, να συνεχίσει το έργο μας για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, να συνεχίσει να προστατεύει τα θύματα των εγκληματικών πράξεων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσπάθειες που έχετε κάνει στο πλαίσιο του κανονισμού για την καταπολέμηση της παιδικής πορνογραφίας, της σεξουαλικής βίας, των σεξουαλικών εγκλημάτων. Οι λύσεις στις οποίες καταλήξαμε θα προστατεύσουν τα πλέον ευάλωτα θύματα, συγκεκριμένα τα παιδιά. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Αντζελίνη, την εισηγήτρια, για τις ε, προσπάθειές της. Έδειξε αξιοθαύμαστη αφοσίωση χάρη στην οποία ηγήθηκε όλων των προσπαθειών ε, που έγιναν ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Έστεφθη με επιτυχία το εγχείρημά της, ε, διότι με ομοφωνία σχεδόν υπερψηφίστηκε το σχέδιό της, αφού, αφού λύσαμε το μεγάλο πρόβλημα των πίνακων συσχετισμών των πινάκων σχετισμών. Το σχέδιο επίσης θα σταλεί προς υπογραφή την ερχόμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, προστατεύουμε και πάλι εδώ τα θύματα ε, των αξιόπινων πράξεων και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες παρά τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίσουμε. Επίσης, υπάρχει ο κανονισμός για το δικαίωμα ενημέρωσης ε, σε θέματα ποινικού δικαίου. Το θέμα αυτό θα ψηφιστεί στις 12 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια και ελπίζουμε ότι θα γίνει αποδεκτό και αυτό στην μετά την πρώτη ανάγνωση. Η Πολωνική Προεδρία επίσης δρομολόγησε τις εργασίες σχετικά με το σχέδιο οδηγίας για τη θέσπιση ελαχίστων προτύπων για την προστασία των θυμάτων αξιόπινων πράξεων. Η Πολωνική Προεδρία ε, διοργάνωσε ένα διάλογο όπου συμμετείχαν εθνικοί εμπειρογνώμονες ο στόχος είναι ε, να χορηγηθεί ε, προστασία στα θύματα όταν υπάρχει σωματική βία. Μιλήσαμε για την απομάκρυνση των θυμάτων από τους δράστες, ειδική προστασία για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες θυμάτων. Ελπίζουμε ότι στη σύνοδο του Δεκεμβρίου θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε το υποσυζήτηση σχέδιο ή τουλάχιστον εν μέρη για να το διαβάσουμε στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για το ενδιαφέρον που δείχνει και τις προσπάθειες που κάνει σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης. Το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη προβήκαμε σε ανταλλαγή απόψεων με τους εισηγητές. Ελπίζουμε ότι την επόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο θα μπορέσουμε τουλάχιστον να εγκρίνουμε μια ε, μητελή κοινή προσέγγιση για το σχέδιο που συζητούμε. Σας ευχαριστούμε πάντως για τις προσπάθειες που κάνατε για το σχέδιο ε, οδηγίας για το δικαίωμα ε, ε, για δικαστική, δικηγορική υπεράσπιση. πρόκειται για το τμήμα Γ της ε, οδηγίας, καταφέραμε παρά τα προβλήματα να πλησιάσουμε περισσότερο μία συμβαστική λύση. Αληθεύει ότι εκκρεμούν πολλά ζητήματα για τα οποία χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. Ε, επίσης, στη Βαρσοβία διοργανώσαμε μία διήμερη διάσκεψη για την ε, ε, υποστήριξη εξοφίκιο των θυμάτων των αξιόπινων πράξεων από κοινού με την, ε, τον Ευρωπαϊκό Σύλλογο Δικηγόρων στην Τρίρ, στην Γερμανία. Ένα μέλος της Επιτροπής η κυρία Αντωνέσκου συγκεκριμένα. Η κυρία Αντωνέσκου, λοιπόν είναι η συγγήτρια για αυτό το θέμα και θα έρθω σε επαφή μαζί της ε, αύριο στην ε, διάσκεψη. Θα θέλαμε στην, ε, στο επόμενο Συμβούλιο να παρουσιάσουμε τις συμβαστικές λύσεις που θα έχουμε καταλήξει στην εργασία με τα κράτη-μέλη για να μπορέσει η Ιδανική Προεδρία να συνεχίσει το έργο μας και να ολοκληρώσει τις προσπάθειές μας. Επίσης έχουμε στείλει στις ομάδες εργασίας ε, σχέδια σχετικά με τα περιουσιακά ε, στοιχεία, τα γαμικά περιουσιακά στοιχεία, έχουμε εντοπίσει ήδη τα προβληματικά σημεία που πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω στις ε, ομάδες εργασίας των εμπειρογνωμών για τα ζητήματα αυτά. Ελπίζω να καταδείξαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα πολιτικό κατασκεύασμα, δεν είναι μόνο για πολιτικούς, Βοηθάει και τους πολίτες να ε, λύνουν τα καθημερινά τους προβλήματα, όπως αυτά που προανέφερα. Και θα ήθελα ακόμη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε. καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Σας διαβεβαιώ ότι θα συνεργαστούμε στενά με τις δύο επερχόμενες Προεδρίες για αυτά τα ζητήματα και παραμένω στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Τσιάλουκ, έχουμε μάθει όλοι πολωνικά από τον πρόεδρό μας, τον κύριο Ζέζι Μπούζεκ. Έχουμε Νομίζω πολλά θέματα να συζητήσουμε. Ήδη κάποια μέλη της Επιτροπής έχουν ζητήσει το λόγο για να υποβάλουν ερωτήσεις. Ε, σίγουρα θα έχετε και χρόνο για να μας απαντήσετε. Η κυρία Κόντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Πολωνική Προεδρία με χαροποίησε το γεγονός ότι συνεχίζεται το έργο της Ουγγρικής Προεδρίας, όπως είπατε στην παρουσίασή σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Μία ερώτηση για την ε, προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ε, ζώνη Σέγγεν. Ξέρετε ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι αξιόπιστη. Ε, θα ήθελα να ξέρω πώς βλέπετε να εξελίσσετε η διαδικασία, πώς ε, θεωρείτε ότι μπορείτε να βοηθήσετε τη διαδικασία αφενός. Αφετέρου, υπήρχε μια σαφής δέσμευση να προχωρήσει το θέμα του ασύλου και το Κοινοβούλιο ήθελε να έχει αυτό το θέμα του ασύλου από κοινού ευθύ εξ αρχή. Τώρα βλέπουμε όμως ότι κάποια πράγματα προχωρούν ενώ κάποια άλλα έχουν κολλήσει στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την άποψή σας για το ε, κατά πόσον μπορείτε να βοηθήσετε αυτή τη διαδικασία. Επίσης είπατε ότι θα παρακολουθήσετε τις διαπραγματεύσεις ε, για τη Συμφωνία για την Προστασία Δεδομένων με τις ΗΠΑ. Θα ήθελα να μάθω κάποια περισσότερα πράγματα και από εσά να ε, μας πείτε λίγα περισσότερα για τη διαδικασία και να μας πείτε και πώς το βλέπετε, ε, διότι γνωρίζετε κι εσείς υπάρχουν διαφορές ερμηνείας ε, στα θέματα της προστασίας δεδομένων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπουσουτήλ, ε, έχετε ζητήσει το λόγο συντονιστές του ΕΛΚ και τον λαμβάνετε φυσικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ξεκινήσω με μια διευκρίνηση. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα ε, θέτουμε ερωτήσεις για τα θέματα δικαιοσύνης, έτσι, όχι για τα θέματα ιστορικών υποθέσεων. Ωραία. Θα έχουμε και τη δυνατότητα να θέσουμε και αυτά τα ζητήματα αργότερα. Ο πρόεδρος μιλάει εκτός μικροφώνου. Ωραία, θα σταθώ στις, ε, στον πρώτο μιλητή. Κάποια θετικά πράγματα έχω να πω. Εξ ονόματος του ΕΛΚ θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας, αλλά κατά δεύτερον, το πιο σημαντικό, να σας ευχαριστήσω για τα όσα κάνετε σε τόσους πολλούς τομείς και ιδίως στο νέο και συναρπαστικό τομέα του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Έγινε πολύ σημαντική πρόοδος στο θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Προστασίας, μόλις το ψηφίσαμε άλλωστε, και αναφερθήκατε κι εσείς στη νέα νομοθεσία για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και το δικαίωμα στην ενημέρωση σε ποινικά ζητήματα. Επιπλέον ε, ευχαριστούμε την Πολωνική Προεδρία διότι ξεκίνησε τις συζητήσεις για νέες προτάσεις όπως για παράδειγμα ε, τα θύματα ε, ποινικών αξιόπινων πράξεων, φαντάζομαι ότι η συνάδελφος θα σχολιάσει, και το δικαίωμα σε δικηγόρο. κύριε Υπουργέ, εμείς θεωρούμε ότι σε αυτό το νέο τομέα δεν αναφερόμαστε απλώς και μόνο σε ένα νέο τομέα, αναφερόμαστε σε ένα νέο τρόπο ε, λήψης αποφάσεων και μεθοδολογίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας έχει πλέον ε, πλήρη εξουσία και δικαίωμα συναπόφασης με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η συνεισφορά του ε, Κοινοβουλίου θα μας οδηγήσει σε πιο ποιοτικέ αποφάσεις, οι οποίες θα μας οδηγήσουν με τη σειρά τους σε καλύτερη νομοθεσία και θα αυξήσουν τα δικαιώματα των πολιτών, διότι θεωρούμε ότι το επόμενο πιο σημαντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την ενιαία αγοράς είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, στον οποίο οι πολίτες μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα, με την εγγύηση ότι θα έχουν την ίδια πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο στα λόγια. Ε, στην πράξη, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπάρχουν ακόμα εθνικά σύνορα σε θέματα ποινικού δικαίου, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Οι πολίτες εξακολουθούν να φοβούνται να μετακινηθούν, διότι φοβούνται την έλλειψη προστασίας σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για όλα όσα κάνατε. Σα υποστήριξε η ομάδα του ΕΛΚ σε όλα όσα κάνατε. Τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα άλλωστε είχαν οι συγητές του ΕΛΚ και θα ήθελα να σα συγχαρώ για το έργο σα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητά το λόγο. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο τώρα. Από τους φιλελευθέρους δεν είχαμε κανέναν. Ευχαριστώ. Μπερδεύτηκα λίγο γιατί νόμιζα ότι θα τα συζητήσουμε όλα μαζί. Θα σταθώ λοιπόν μόνο στα θέματα δικαιοσύνης. Έχω την εξής παρατήρηση. Ο Υπουργός μας είπε ότι η συζήτηση για την ε, πρόσβαση σε δικηγόρο είναι ακαθόδες ζήτημα, αλλά έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδο. Συμφωνώ, είναι ακαθόδεστο ζήτημα, αλλά δεν διαβλέπω κάποια πρόοδο, διότι φαίνεται ότι και οι Δανείοι συνάδελφοί σα που θα αναλάβουν τα ενία δεν θεωρούν ότι το θέμα του δικαιώματο σε δικηγόρο αποτελεί προτεραιότητα για το δικό του εξάμεινο. Και αυτό μα οδηγεί στη μεγαλύτερη συζήτηση, που είναι το θέμα τη αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ε, η ευρωπαϊκή συνεργασία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και ότι το θέμα της αμοιβέ εμπιστοσύνης δεν είναι πάντα υγιές, διότι ορισμένες φορές τα σοφρονιστικά καταστήματα σε κάποιες χώρες δεν είναι εξίσου καλά με άλλα και λίγα σας λέω και η αμοιβέ εμπιστοσύνη βεβαίως δεν είναι πάντα τόσο καλή αν δούμε ότι τα ευρωπαϊκά ένταλμα σύλληψη οδηγεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πολίτε οι οποίοι αποστέλλονται από τη μία χώρα στην άλλη για ε, μακροπρόθεσμη προδικαστική κράτηση για ένα ε, αδίκημα τα οποία είτε δεν διέπραξαν είτε ε, δεν ε, είναι στα δικήματα τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία της τόσο μεγάλης προδικαστικής διαδικασίας. Είπατε ότι η χώρα σας χρησιμοποιεί πολύ το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, Σύλληψης. Έχω δει τα ποσοστά να πέφτουν, αλλά εξακολουθείτε να είστε ε, πρώτοι και να έχετε τα πρωτεία στο θέμα αυτό. Θεωρείτε ότι αν είχε ξεκινήσει η συζήτηση για τη σωστή χρήση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ε, Σύλληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης ε, θα έπρεπε ίσως να ξεκινήσει, διότι νομίζω ότι οι πολίτες μας δεν απολαμβάνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη όταν ε, βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης και τους αποστέλλεται ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για μια ε, σύλληψη σε άλλη χώρα. Η κυρία Μποσκούρ. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση. Ξέρω ότι έχουμε κάποιον που εκπροσωπεί εδώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά θα πρέπει να κάνω την ερώτησή μου παρόλα αυτά, γιατί αλλιώ κανείς δεν θα μου απαντήσει. Όσον αφορά την έλλειψη διακρίσεων και παρόλο που η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά, δεν ήρθε εδώ ποτέ αρμόδιος υπουργός ε, για τα θέματα αυτά. Αφού λοιπόν εσείς είστε εδώ σήμερα, θα ήθελα να μου πείτε όσον αφορά την οδηγία για τις διακρίσεις, ποια είναι τα θέματα τα οποία θα δώσετε στους Δανούς στην επόμενη Προεδρία. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πολλά πράγματα δεν προχωρούν και ότι θα πρέπει να προσφέρουμε καλύτερη προστασία στους πολίτες της Ευρώπης τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν στην καρδιά της Πολωνικής Προεδρίας. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι κάνετε για το θέμα αυτό. Όσον αφορά τώρα την πορνογραφία, τη βία με θύματα τα παιδιά. Η τροπολογία μου υιοθετήθηκε και πρόκειται για θέμα ποινικού μητρώου. Αυτό πιστεύω ότι σίγουρα θα βελτιώσει την κατάσταση, αλλά είναι πολύ σημαντικό εφόσον κάποιος καταδικαστεί και αφού τελειώσει η περίοδος φυλάκισης του να μην μπορεί να ξαναεργαστεί με παιδιά, να υπάρχει η καταδίκη του και ο, και ο λόγος στο ποινικό μητρό το οποίο θα τον ακολουθεί. Ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε. Θα γίνει το πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Πολωνία του χρόνου. Οι απάτες στον αθλητισμό είναι κάτι που σίγουρα μας απασχολεί και που σίγουρα εμπίπτει στην συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού Ξέρω ότι εδώ χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ των Υπουργών, των Υπουργείων Αθλητισμού, αλλά και των αστυνομικών αρχών και είναι θέμα αρμοδιότητας του Υπουργού Δικαιοσύνης. Πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα, πολλές φορές με διεθνείς διαστάσεις και βλέπουμε ότι υπάρχουν και στενές διασυνδέσεις με τη λεύκανση βρωμικού χρήματος, με τα ναρκωτικά και με την τρομοκρατία. Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι πρόκειται για εγκλήματα τα οποία πολλές φορές δεν απασχολούν αρκετά τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, όσον αφορά την τρομοκρατία, είδαμε ότι ο Ισλαμισμός απασχολεί ιδιαίτερα τις αρχές και πολύ λιγότερο τα εξτρεμιστικά κινήματα όπως αυτά που σήμερα εμφανίζονται στην Γερμανία. Ακροδεξιά ακραία κινήματα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ιδιαίτερα το τι γίνεται στη Γερμανία και σε άλλες χώρες με τον ακροδεξιό αυτόν εξτρεμισμό. Κυρία Χιμένες Πεχερίλη, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, Υπουργό εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας, διότι μας ε, βοήθησε και έδωσε όθηση για το νόμο για την προστασία των θυμάτων. Ήταν ε, υποδειγματική η Προεδρία σε όλα τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των θυμάτων και θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ερώτηση στο ίδιο θέμα, διότι εγώ είμαι η για το δικαίωμα στην προστασία των θυμάτων, ε, θύματα ε, εγκληματικών πράξεων, τα οποία συζητάμε τώρα και τα οποία γνωρίζω ε, ότι ω ζήτημα απασχόλησαν ιδιαίτερα την Πολωνική Προεδρία και τα υποστήριξε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, όταν τέθηκε το θέμα της προστασίας των θυμάτων, όλοι ε, καλωσόρισαν αυτό το ζήτημα, αλλά αυτή η αρχική ψευδέστηση άρχισε να χάνει ε, λίγο την έγκλη της, διότι άρχισαν να συζητούν για περιορισμούς ε, στο Συμβούλιο. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να το περιορίσουμε. Ίσα ίσα θέλουμε να το διευρύνουμε κατά πολύ και ελπίζω ότι με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το νομοθετικό αυτό το κείμενο και όχι να το περιορίσουμε. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι άποψη έχετε εσείς Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να δώσουμε μία όθηση στη Δανική Προεδρία ε, εάν θα δώσουν και αυτή τη μάχη μας ή δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Πώς θεωρείτε ότι μπορούμε να προωθήσουμε το θέμα της προστασίας των θυμάτων ε, και να συμπεριλάβουμε και τα θύματα τρομοκρατίας, τα θύματα οργανωμένου εγκλήματος, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι είναι βάλλοντες ομάδες, υπάρχει θέματα ανηλίκων, ε, θέματα εμπορίας ανθρώπων, ε, ε, βία κατά των γυναικών και να υπάρχει η νομοθεσία αυτή η οποία πρέπει να υπάρχει για να μπορούν να προστατεύονται τα θύματα και οι οικογένειές τους και ταυτόχρονα να υπάρχει και συνδρομή σε ψυχολογικό επίπεδο, δικαίωμα στη διερμηνία, πράγματα τα οποία συνήθως προσφέρονται ε, στους θήτες αλλά για κάποιο κατανόητο λόγο είναι ε, κάτι το οποίο δεν διαθέτουν τα θύματα. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό, ώστε η επόμενη Προεδρία να κάνει ό,τι έκανε και αυτή η Προεδρία, να προχωρήσει το θέμα ε, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Προστασίας και να εγκριθεί. θεωρείτε ότι με τη βοήθειά σας μπορούμε να δώσουμε μια όθηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ρομέρο Λόπεθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, επειδή ήμουν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας, για τις γυναίκες ε, θύματα βίας, να Από τι φορά τιμή στην Πολωνική Προεδρία, διότι έκανε τεράστιες προσπάθειες να υλοποιηθεί αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα προστασίας. Αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί θα ήταν να μην το θεωρήσετε προτεραιότητα και από εκεί και πέρα θα έπρεπε να περιμένουμε την Προεδρία της Δανίας, όπως έγινε και στο παρελθόν σε κάποιε περιπτώσει. Αυτά όλα όμως ε, τα προώθησε η Πολωνική Προεδρία και έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Όσον αφορά τις δικαστικές διαδικασίες, θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπατε για το... θέμα της πρόσβασης σε νομική συνδρομή, ε, πρόσβαση σε δικηγόρο και τη σχετική οδηγία. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στην περίπτωση ε, που ο ύποπτος έχει δικαίωμα στο δικηγόρο, αλλά το να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε χώρα μέλος και τι δισταγμοί υπάρχουν, ποια είναι τα κράτη-μέλη τα οποία ε, υποβάλλουν περισσότερες ε, προτάσεις, ποιοι έχουν περισσότερες δισταγμούς. Να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης για να ξέρουμε και τι θα γίνει με την Εδανική Προεδρία. Όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για το άσυλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις μας παρουσίασε ένα έγγραφο και αυτό που ισχύει είναι ότι στο έγγραφο δεν διευκρινίζεται τίποτα για τις προτάσεις που έκανε η Πολωνική Προεδρία για την τροποποίηση του κανονισμού Δουβλίνου. Θα ήθελα να ξέρω τι προβλήματα υπήρχαν, τι προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται για την ε, τροποποίηση του κανονισμού του Δουβλίνου και τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσει η Δανική Προεδρία για το θέμα αυτό και κάτι το οποίο σχετίζεται και με αυτό που συζητάμε, τι στάση τήρησε η Πολωνική Προεδρία και τι στάση μπορεί να τηρήσει η Δανική Προεδρία για το θέμα της ε, τροποποίησης των συνόρων ε, στη ζώνη Σέγγεν. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός τώρα θα απαντήσει. Να σας υπενθυμίσω ότι είναι εδώ και οι δύο εκπρόσωποι της Πολωνικής Προεδρίας και ο κύριος Τζάλου και ο κύριος Σάνσκικ. Και νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματος όλης της Επιτροπής όταν αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο προέδρευσε η Πολωνική Προεδρία στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Τα πιο ουσιαστικά ζητήματα νομίζω ότι πραγματικά μπορέσετε να συνεισφέρετε και θα ήθελα αυτό να καταγραφεί. Έχετε το λόγο, Υπουργέ. Dziękuję bardzo ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ ιδιαίτερα διότι αναγνωρίσατε αυτά που πέτυχε η Πολωνική Προεδρία. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε εξαιρετική συνεργασία και πολύ εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ της Πολωνικής Προεδρίας και της Επιτροπής σας. Όντως, την καρδιά αυτών που θέλησαμε να κάνουμε είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά τις ερωτήσεις τώρα που μου κάνατε, εντοπίσατε τις ερωτήσεις σας εν μέρη σε θέματα που δεν είναι της αρμοδιότητας ε, του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όσον αφορά την ε, του Δουβλίνου και αυτές που αφορούν το άσυλο, τις σημείωσα και ο Υπουργός Ταχάντζεκ θα δώσει απαντήσεις σε αυτές. Κύριε Μπουσούτιλ, έχετε δίκιο. Όντως, εργαζόμαστε προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει με ένα νέο κείμενο, νέα συνθήκη, νέο σύστημα εξουσιών και αρμοδιοτήτων από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και βεβαίως αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εργάστηκε η Πολωνική Προεδρία. Επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη φορά που προεδρεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε λοιπόν εμπειρία και δεχτήκαμε την συνθήκη της Λισαβόνας σαν την νομική υποδομή μας στην οποία πρέπει να λειτουργήσουμε. Έγινε ένας μεγάλος αριθμός ε, συνεδριάσεων με συμμετοχή των ε, εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο τρίλογος, η συζήτηση που έγινε, νομίζω ότι έδειξε ότι υπάρχει ανοιχτό πνεύμα και ότι είμαστε διατεθειμένοι, ήμασταν διατεθειμένοι να δεχτούμε το ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει των συνθήκων. Είναι επίσης σαφές ότι πραγματικά βασιστήκαμε στην εμπειρία μας από την χώρα μας. Σε μας το Κοινοβούλιο είναι εξαιρετικά ισχυρό. Δεν ξέρω αν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στα πρότυπα και στις απαιτήσεις της συνθήκης της Λισαβόνας. Παρ' όλα αυτά κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ό,τι καλύτερο μπορούσαμε έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι όπως ε, αναφέρει και η συνθήκη, οι δύο νομοθετικές αρχές αντιμετωπίζονται επίσης όρις όσον αφορά την νομοθετική εργασία. Επίσης υπήρχαν και κάποιες ερωτήσεις που αφορούσαν την οδηγία για θύματα εγκλημάτων. Ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωμα σε υπεράσπιση, η προστασία των θυμάτων. Νομίζω ότι καταρχήν μπορώ να πω ότι το σχέδιο της οδηγίας έγινε γνωστό στο τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας. Άρα όλες οι συζητήσεις έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο έγγραφο που απορρέει από προηγούμενες αποφάσεις, είναι το αποτέλεσμα προηγούμενων αποφάσεων πάνω στις οποίες βασιστήκαμε. Υπάρχουν επίσης και κάποιες αξιολογήσεις οι οποίες αφορούν το πλαίσιο στο οποίο έγινε όλη αυτή η εργασία. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είχαμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Σημειώστε όμως ότι έγινε πολύ σημαντική πρόοδος για το θέμα αυτό. Όπως είπα και στα εισαγωγικά μου σχόλια, μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε έναν μεγάλο αριθμό θεμάτων. Κάποιες άλλες έχουν προχωρήσει σημαντικά, όπως παραδείγματο χάρη το θέμα της εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Πιστεύω λοιπόν ότι η επόμενη Προεδρία, η Δανία, θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τα υπόλοιπα θέματα. Αναφέρθηκα λοιπόν στην συνέχεια της εργασίας ε, της προηγούμενης προεδρίας, της Ουγγρικής Προεδρίας. Πρέπει να σας πω ότι η δική μου αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεργασία μας με την Ουγγαρία ήταν εξαιρετική. Εν πάση περιπτώσει, συνεργαστήκαμε εξαιρετικά από την αρχή της Προεδρίας μας με την Ουγγρική Προεδρία. Και βεβαίως ε, προετοιμάσαμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο τηρήσαμε χωρίς βιασύνες και χωρίς παραλήψεις. Συνεχίσαμε λοιπόν τις ε, εργασίες της Ουγγρικής Προεδρίας και αξιολογώντας αν θέλετε τον αριθμό των ε, νομοθετικών εργασιών που ολοκληρώσαμε, διαπιστώσαμε ότι αυτό δεν είναι το μόνο κριτήριο για την επιτυχία μιας προεδρίας. Ιδιαίτερα αν κανείς δει τη σημασία που έχει ένα θέμα όπως η προστασία των θυμάτων εγκληματικής δραστηριότητας. Ελπίζουμε εδώ η Δανέζικη Προεδρία να ολοκληρώσει τα θέματα που παραμένουν εκρεμή. Δεν πρέπει να κλείσουμε με βιασύνη τόσο σοβαρά θέματα, γιατί αν λάβουμε κάποιες αποφάσεις βεβιασμένα, αυτό μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα. Πολλά θέματα μας φάνηκαν πολύ πιο απλά στην αρχή, αποδείχτηκαν πολύ πιο περίπλοκα. Και αυτό για πολλούς λόγους. Παραδείγματος χάρη, είμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όπου η οικονομική κρίση δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ τα πράγματα. Τα θύματα εγκλημάτων, η πρόσβαση στην υπεράσπιση κάτι το οποίο χρηματοδοτούν τα κράτη βεβαίως, σαφώς και προϋποθέτουν χρηματοδότηση από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Η θέση λοιπόν της Πολωνικής Προεδρίας ήταν ε, από την αρχή να θεωρήσει ότι δεν είναι δυνατόν να υιοθετηθούν λύσεις οι οποίες είναι δίκαιες και δεν έχουν καμία οικονομική επίπτωση. Κάποιος θα πρέπει να αναλάβει το κόστος αυτής της υπεράσπισης παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό και είμαστε πολύ πιο συντηρητικοί αν θέλετε στις διαπραγματεύσεις μας. Εμείς όταν συζητούμε τέτοια θέματα στη χώρα μας έχουμε πάντα τον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Οικονομικών ο οποίος μας προσγειώνει αν θέλετε. Και μετά από μια ολόκληρη σειρά αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά συγκεκριμένα την πρόσβαση ε, στην υπεράσπιση. Αναφέρομαι εδώ σε πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Συνειδητοποιούμε ότι Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί εκτενώς ε, στην Ευρώπη και πολλές από τις ε, αποφάσεις αυτές ε, του δικαστηρίου είναι αποφάσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Βλέπουμε όμως ότι τα κράτη-μέλη, πολλά κράτη-μέλη, αντιδρούν, διστάζουν να προχωρήσουν στις απαραίτητες αυτές αλλαγές για να μπορέσουν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις. Ήμασταν λοιπόν ίσως πολύ φιλόδοξοι, η Πολωνική Προεδρία ήταν πολύ φιλόδοξη και δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει όλα αυτά τα τόσο φιλόδοξα σχέδια. Ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία στη Δανέζικη Προεδρία και σε έξι μήνες ελπίζουμε τα νέα να είναι καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών. Η κυρία Σαργεντίνη αναφέρθηκε σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα για την Πολωνία. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε μία διμερή συζήτηση αργότερα Χαίρομαι ιδιαίτερα πάντως γιατί διαπιστώσατε ότι ο αριθμός των ενταλμάτων στην Πολωνία είναι πολύ σημαντικός παρόλο που μειώνονται. Είμαστε, αν θέλετε, στην περιοχή μας η μεγαλύτερη χώρα και ίσως είναι λογικό σε απόλυτους αριθμούς να είμαστε και πρώτοι. Σε αριθμούς πάντα. Πέρσι είδαμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο επεξεργάστηκαν το θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Εμείς ε, θέλουμε να υποβάλουμε το θέμα αυτό στην επόμενη συνάντηση του Συμβουλίου και στο κείμενο που έχουμε προετοιμάσει προτείνουμε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ένταλμα. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών και ενδεχομένω αυτό να οφείλεται και στο γεγονό ότι κάποιε αποφάσει πλαίσιο έχουν ληφθεί κάπω βεβιασμένα. Σε μια συγκεκριμένη πολιτική κατάσταση που βρισκόταν ε, τότε η Ευρώπη. Η Προεδρία βεβαίως και έχει σημειώσει και τη συζήτηση που συνεχίζεται όσον αφορά την αναρμόνιση των συνθήκων παραμονής ε, σε κέντρα κράτησης, το χρόνο, τις συνθήκες. Η συζήτηση για τα θέματα αυτά συνεχίζεται, βρίσκεται εν εξελίξη και την ίδια ώρα διαπιστώνουμε ότι τα κέντρα κράτησης μπορεί πραγματικά να επηρεάσουν τις εφαρμοσκές διατάξεις του εντάλματος σύλληψης, του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως θα είχαμε αρχικά όπως τα είχαμε αρχικά τουλάχιστον εκτιμήσει. Υπάρχουν κάποια εθνικά ή περιφερειακά χαρακτηριστικά θα έλεγα που πραγματικά επηρεάζουν αυτό το εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως, ίσως και οι πιο σκληροί να έχουν κάπως μετριάσει αυτή τη στιγμή την στάση τους και η πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση είναι κάτι που θα επικρατήσει όπως παραδείγματο χάρη οι αναφορές του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ε, ανθρώπινη αντιμετώπιση των κρατουμένων, την απαγόρευση των βασανιστήριων και βεβαίως εδώ γίνεται και μια σαφής αναφορά στην Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ίσως αυτά τα κείμενα δεν ε, έχουν ε, κυρωθεί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και το σύστημα δεν λειτουργεί ομοιογενώς και πολλές φορές βλέπουμε ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν ε, υλοποιούνται και δεν εφαρμόζονται πάντα. Η Πολωνική Προεδρία βεβαίω δεν μπόρεσε να ανοίξει το θέμα αυτό καθότι υπάρχουν κράτη-μέλη που αντιδρούν. Η Πολωνία είναι διατεθειμένη πάντω να προχωρήσει σε επεξεργασία και συζήτηση για το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Μπόσκοβιτς για την οδηγία για τις διακρίσεις, την αποφυγή των διακρίσεων. Όντως δεν είναι αυτό θέμα δικής μου αρμοδιότητα. Η Πολωνική Προεδρία, από ό,τι ξέρω, έχει ολοκληρώσει την εργασία αυτή προετοιμάζοντας και υποβάλλοντας μία έκθεση προόδου όσον αφορά την ηλικία, τις διακρίσεις βάσει της ηλικίας και πιστεύω ότι η εργασία αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Δανίας. Από ό,τι φαίνεται, ο παράγοντας ηλικία αποτελεί έναν τρόπο για να συνεχίζονται οι διακρίσεις. Οι νέοι αλλά και οι πιο ηλικιωμένοι είναι <coughs> θύματα διακρίσεων. Τώρα, όσον αφορά την τροπολογία για την σεξουαλική κακομεταχείριση των παιδιών, και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και όσον αφορά τους ποινικού κώδικες των διαφόρων χωρών. Το θέμα αυτό, όπως ξέρετε, μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα. Υπάρχει βεβαίως η περίφημη υπόθεση Dutroux, από την οποία ξεκίνησε η αναρμόνιση των ε, ευρωπαϊκών νομοθεσιών για τα θέματα αυτά. και το θέμα βεβαίως των κυρώσεων και βεβαίως την αποφυγή δυνατότητας να ξαναεργαστεί κανείς με παιδιά αφού ολοκληρώσει την φυλάκισή του. Αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνω όμως θα συνεχιστεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί από την Πολωνική Προεδρία και ενδεχομένως συμφωνώ μαζί σας ότι το θέμα αυτό δεν αποτέλεσε προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρόλες τις προσπάθειες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εδώ το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Όσον αφορά την νομοθεσία της Πολωνίας, νομοθεσία κατά της διαφθοράς, γιατί την καταπολέμηση της διαφθοράς, Έχουμε τέτοια νομοθεσία στη χώρα μας. Το πόσο βέβαια αποτελεσματική είναι αυτή η νομοθεσία στην Πολωνία αλλά και αλλού όσον αφορά την πρόληψη τέτοιας εγκληματικής δραστηριότητας που όντως είναι μια δραστηριότητα που γεννά ενδιαφέρον γιατί είναι εξαιρετικά κερδοφόρα. Μιλήσατε για τις απάτες στον τομέα του αθλητισμού και αυτό το θέμα θα πρέπει σαφώς να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας από τις επόμενες προεδρίες, τη Δανέζικη Προεδρία. συμφωνώ και με τις ε, δύο τελευταίες παρατηρήσεις των Ισπανών συναδέλφων που μίλησαν ε, για την υπεράσπιση. Είναι πάρα πολύ, αν θέλετε, εντυπωσιακό να δει κανείς το πόσο διαφορετικές λύσεις προτείνουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά το θέμα αυτό της υπεράσπισης και της πρόσβασης ε, σε δικηγόρο. Οι λύσεις είναι πάρα πολύ διαφορετικές από τη μια χώρα στην άλλη και η Πολωνική Προεδρία ξεκίνησε διαπραγματεύσεις ε, για το θέμα αυτό και προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών από τη μία και την ε, διαδικασία και την σωστή λειτουργία της δικαιοσύνης από την άλλη. Διότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμποδίσουμε τις δικαστικές αρχές να προχωρήσουν στην διερεύνηση μιας υπόθεσης. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχουν προβλήματα και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί πολλές φορές για λόγους διαδικαστικούς οι αρχές υποχρεούντα να απαγορεύσουν την πρόσβαση των δικηγόρων για διαδικαστικούς λόγους και πολλές φορές αυτό είναι απαραίτητο αλλά αυτό πρέπει να γίνεται όσο είναι απαραίτητο για την ορθή λειτουργία δικαιοσύνη και όχι παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να μην έχετε πλέον αμφιβολίες και ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε κυρία Τζιάλουκ. Εκτιμούμε τις προσπάθειες που κάνετε για να απαντήσετε διεξοδικότατα σε όλες τις ερωτήσεις. Ε, όντως δώσατε λεπτομερείς απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που ήγηραν οι βουλευτές. Η κυρία Μπότσκουρτ όμως βλέπω θέλει να κάνει μια επερώτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό που μου έδωσε μια λεπτομερή απάντηση. Υπάρχει όμως κάτι στο οποίο δεν απαντήσατε. Σε ποιο βαθμό λαμβάνουμε υπόψη ε, την ανάγκη καταπολέμησης ε, της ε, ακροδεξίας, δηλαδή συνιστά προτεραιότητα τελικά για την Ένωση η καταπολέμηση ανώδου της ακροδεξίας. Απάντηση. Είναι όντως ε, ένα νέο ζήτημα που μας απασχολεί. Ε, υπάρχουν πολλές νέες απειλές. Ε, σας θυμίζω τι συνέβη στην Νορβηγία την επίθεση που ε, έλαβε χώρα στο νησί της Νορβηγίας ε, κατά των ε, εκδηλωτών. Ουσιαστικά θα πρέπει να συμφωνήσουμε αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις αξιόπινες πράξεις που διαπράττουν αυτά τα ακροδεξιά κινήματα. Δηλαδή, σε ποια κατηγορία θα πρέπει να ενταχθούν. Η εγκληματολογία δεν είμαι σίγουρος ότι θα και ικανοποιητικά επιχειρήματα ώστε να ανακηρύξει τα ακροδεξιά κινήματα σε, αν θέλετε, πιο επικίνδυνους εχθρούς σε σχέση με άλλα ρισοπαστικά ακραία κινήματα. Δεν ε, κρίναμε ότι ήταν ε, επιτακτική η ανάγκη να χειριστούμε ξεχωριστά αυτό το ζήτημα. Όντω συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας, αλλά το θέμα της ε, αυξημένης βίας που προέρχεται όμως από όλων των ειδών τα ριζοσπαστικά κινήματα είναι μια απειλή ε, που θα έπρεπε να καταπολεμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να γίνει πρώτα διάλογο σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι μετά τις ερωταπαντήσεις μπορούμε να ακούσουμε και τη δεύτερη παρουσίαση του κύριου Πιότρε Σταχάνσης. Ε, συγγνώμη, το παρεύθυρα φαντάζομαι. χαρήκαμε ιδιαίτερως που λάβαμε τόσες πολλές απαντήσεις για τα θέματα δικαιοσύνης. Σας περάσουμε τώρα ε, στο τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Εσωτερικών υποθέσεων, έχετε το λόγο. Κύριε Σταχάντζιτς, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω το έργο της Πολωνικής Προεδρίας στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων. Αναμφισβήτητα, το στοιχείο κλειδί που συνιστά και προτεραιότητα για την Προεδρία μας ήταν ό,τι σχετίζεται με το σύστημα χορήγησης ασύλου στην Ένωση. Ο στόχος της Προεδρίας ήταν να αναλυφθεί κάθε πιθανή δράση ώστε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που είχε προκαθοριστεί, ε, δηλαδή το τέλος του 2012, για την θέσπιση του νέου συστήματος. Γνωρίζετε πολύ καλά βεβαίως πως το νομικό πακέτο που ονομάζεται κοινοτικό πακέτο ασύλου απαρτίζεται από πέντε νομοθετήματα. Ως προς την οδηγία ε, χαρακτηρισμού κάποιου, δηλαδή Qualification Directive, Σημειώθηκε πρόοδο ε, για το περιεχόμενο του σχεδίου και χάρη στη συμβαστική λύση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για του πίνακε αντιστοίχηση ε, μπορέσαμε τελικά να προβούμε στην έγκριση του σχεδίου κατά τη διάρκεια τη προεδρία μα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που περατώθηκε λοιπόν. ασχοληθήκαμε όλος ιδιαίτερος με ό,τι σχετίζεται με τις ε, τροποποιήσεις του κανονισμού Δουβλίνου. Στο άτυπο Συμβούλιο Ιστορικών Υποθέσεων Στάπλετ φέτος συζητήθηκε εκτενώς το θέμα και ο στόχος ήταν να ξεφύγουμε από το τέλμα στο οποίο είχε περιέλθει η οδηγία αυτή εδώ και χρόνια. Μπορούμε τώρα να πούμε πως χάρη στις προσπάθειές μας ε, υπάρχει πλέον ένας ε, μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει την αλληλεγγύη με τα κράτη-μέλη που ε, δέχονται μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις. Φασί των συμπερασμάτων ε, του τελευταίου Συμβουλίου που επικύρωσε και η Κορεπέρ στην τελευταία της σύνοδο, αποφασίσαμε να προσθέσουμε νέα ο άρθρο στο κανονισμό του Δουβλίνου ε, για την ε, προεργασία, για την διαχείριση κρίσεων ως προς το άσυλο και για τον το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης. Αυτό το θέμα θα ζητηθεί και την ερχόμενη εβδομάδα στο επόμενο Συμβούλιο Επίσης, στον τελευταίο μήνα της Προεδρίας μας, το Δεκέμβριο, θα επεξεργαστούμε αυτό το θέμα σε επίπεδο ομάδας εργασίας. Ελπίζουμε ότι ε, θα τελεσφορήσει ε, η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα την εισηγήτρια την κυρία Βίξτρομ. Είναι εξαιρετικά καθόδες αυτό το ζήτημα και χαιρόμαστε για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Επίση, ε, κατατέθηκε πρόταση για την ε, ίδρυση ομάδας επαφή. Ε, χάρη λοιπόν σε αυτή την κίνηση της Πολωνικής Προεδρία είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε σχέση με την αποτελμάτωση, όπως σας έλεγα, του κανονισμού Δουβλίνων. Για τον κανονισμό Eurodac για τα δεκτυλικά αποτυπώματα ήταν ένα θέμα που ενδιαφέρε ιδιαίτερα την Πολωνική Προεδρία. Μας ενδιαφέρει ακόμη, ευελπιστούμε ότι θα ε, καταθέσει νέο σχέδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δυστυχώ εμεί εμείς δεν δρομολογήσαμε διαπραγματεύσει. Πρόκειται επίσης για την πρόσβαση στο σύστημα Eurodac. Ελπίζουμε ότι στο άμεσο μέλλον ε, θα σημειωθεί κάποια πρόοδος, ε, διότι Ο στόχο είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλο του 2012 για την οδηγία για την υποδοχή τώρα. Αύριο θα λάβει χώρα η τελευταία συνεδρία της ομάδας εργασίας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη ανάγνωση του σχεδίου και αύριο θα ολοκληρωθούν, ξαναλέω, οι εργασίες της ομάδας εργασίας θα εξακολουθήσουν να υφίστανται διάφορα προβλήματα και πιστεύω ότι η θέση μας θα πρέπει να παραμείνει σαφής. Η Προεδρία της Δανίας ελπίζω να ε, πάρει τη σκητάλη για αυτό το θέμα, διότι έχουμε εργαστεί εντατικά για αυτό το θέμα. Το σχέδιο τώρα για τα διαδικαστικά ζητήματα. Έχουμε επιλύσει κάποια και κυρίως έχουμε εντοπίσει τα βασικά προβλήματα. Ε, η Πολωνική Προεδρία έδωσε περισσότερη βάση στην οδηγία για την υποδοχή. Προσπαθήσαμε όμως να επιλύσουμε προβλήματα και στις υπόλοιπες τέσσερις οδηγίες. Σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Αναφέρθηκα νωρίτερα στο θέμα της αλληλεγγύης, της διακρατικής αλληλεγγύης. Λάβαμε υπόψη αυτή τη συνιστόσα όταν επεξεργαστήκαμε το κανονισμό του Δουβλίνου και Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσει αυτή την άκουσα και η επόμενη Προεδρία. Παραδείγματο χάρη, να συζητηθεί το θέμα του Ταμείου για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες και το άσυλο, συγγνώμη, ε, σχετικά τώρα με την νόμιμη μετανάστευση. πλησιάζουμε στο τέλος ε, των εργασιών μας ε, σχετικά με την κοινή άδεια διαμονής και εργασίας. Η Ουγγρική Προεδρία ήταν μάλλον επιτυχής. Εμείς καταφέρουμε να ρυθμίσουμε αυτό το θέμα του πίνακα ε, αντιστοιχίας. Ε, σχετικά τώρα με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, συμφωνήσαμε επί της πλειοψηφίας των ε, ε, προβλημάτων που είχαν ανακύψει και συμφωνήσαμε επίσης ότι αν δεν εγκριθεί η οδηγία αυτή επί πολιτικής Προεδρίας ε, αναλαμβάνει ταχύτατα να ολοκληρώσει τις εργασίες η επόμενη Προεδρία της Δανίας. Για τους εποχιακούς εργαζομένους τώρα και σχετική οδηγία λύσαμε κάποια προβλήματα, προδέψαμε, αλλά εξακολουθούν να να υπάρχουν μεγάλες διαφορέ από κράτο σε κράτο και θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε αυτό το θέμα. Για τα συνοριακά ζητήματα ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας για την οδηγία για τροποποίηση της εντολής του Frontex. Έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα. Επίση ο Πολωνική Προεδρία τροποποίησε τον κανονισμό για ε, το θύλακα του Καλίνιγκρατ και συγκεκριμένα για την ε, ε, διέλευση των ε, συνόρων. Ελπίζουμε να συνεχιστούν αυτές οι εργασίες. Επίσης, μας απασχολούσαν ε, οι τροποποιήσεις του συνοριακού κώδικα του Σέγγεν. Είχε καταθέσει τεχνικές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις κοινές συνοριακές περιπολίες. Ένα πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας ήταν η ενίσχυση της ζώνης φύλαξης. Η Προεδρία έκανε τις προσπάθειες που χρειάζονταν για να χειριστεί το θέμα, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση οι αλλαγές να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Συζητήσαμε το θέμα του πακέτο διακυβέρνηση του Σέγγεν που δημοσίευσε το Σεπτέμβρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ε, κάναμε την πρώτη ανάγνωση και των δύο ε, σχεδίων του πακέτου, δηλαδή για την αξιολόγηση αποτίμηση του μηχανισμού Σέγγεν, επίσης ε, το σχέδιο για την αξιολόγηση του συνοριακού κώδικα του Σέγγεν. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό μηχανισμό αξιολόγησης και για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος προς τον επιμερισμό των ευθυνών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα επιπροσθέτως η ενίσχυση του συστήματος ε, παρακολούθησης είναι ένα στοιχείο που συνεπάγεται συνέχιση των εργασιών, κυρίως όταν μιλάμε για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των συμβαλωμένων μερών. Ω προ τι ε, αλλαγές, ε, τροποποιήσεις του συνοριακού ε, κώδικα με, με την προσωρινή αποκατάσταση των συνοριακών ελέγχων. Δηλαδή, θυμηθείτε ότι οποιαδήποτε αλλαγή και αν επιφέρουμε δεν μπορεί να παρα, παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και να θέτει εν κινδύνο το την κατοχυρωμένη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να διαχειρίζονται τα σύνορά τους και να παρακολουθούν τις ε, κινήσεις ε, στα σύνορα. Στο επόμενο Συμβούλιο ε, θα συζητηθεί και αυτό το θέμα. Ως προς την καταπολέμηση τώρα του εγκλήματος, το πιο σημαντικό στοιχείο του έργου μας ήταν η καταπολέμηση των εγκληματικών πράξεων σχετίζονται με ναρκωτικά, συνθετικά και μη. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις ανατολικές γειτονικές χώρες για την καταπολέμηση αυτού του είδους των εγκλημάτων και γενικότερα της εγκληματικής δραστηριότητας. Επίσης, Ξεκινήσαμε τις εργασίες για ένα σχέδιο κανονισμού για αυτό το θέμα και ελπίζουμε ότι του χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει σχέδιο για τις ψυχότροπες ουσίες. Ε, τώρα σε σχέση με τα ε, αρχεία δεδομένων και την οδηγία PNR έχουμε προχωρήσει. Οι βασικές αρχές που καθοδήγησαν ε, τις προσπάθειές μας είναι πρώτον η αρχή προστασίας των ατομικών δεδομένων και δεύτερον ε, αρχή διαφύλαξης της διαφάνειας. Ένα τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό θέμα είναι η διεύρυνση της ζώνης του Σέγγεν. Ε, τον Αύγουστο η Πολωνική Προεδρία προετοίμασε ένα σχέδιο συμβαστικής λύσης ε, και έκανε διαπραγματεύσεις ε, για αυτήν την πρόταση όπου συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ε, δυστυχώς το άτυπο εσωτερικών υποθέσεων του Σεπτεμβρίου δεν ενέκρινε τις προτάσεις αυτές. Συνεχίστηκαν παρόλα αυτά οι διαπραγματεύσεις. και αναμένουμε ε, τις ε, δηλώσεις ε, από αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμεί ευχαριστούμε, κύριε Σταχάσνης. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Μπουσούτηλ έχει ζητήσει το λόγο, καταρχάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Υπουργό για την ε, διεξοδικότατη παρουσίαση του έργου της Πολωνικής Προεδρίας για το τόσο ευαίσθητο και διαφιλονικούμενο τομέα που συζητάμε. Να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τον ε, τρόπο με τον οποίο εργάστηκε η Πολωνική Προεδρία στον τομέα αυτό, προχώρησε τα θέματα κατέγραψε μία σειρά από σαφείς επιτυχίες, τις οποίες ε, μας παραθέσετε, δεν χρειάζεται να επαναλάβω εγώ τίποτα. Να πω βέβαια κάτι εν συντομία για τρία ζητήματα. Καταρχάς το θέμα του ασύλου. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ε, μετά από έξι μήνες προεδρία, ότι δεν ε, θα επιλύσουμε το βασικό γρίφο του πακέτου του ασύλου εάν δεν ασχοληθούμε με το θέμα της αλληλεγγύης. Η Πολωνική Προεδρία ήταν πολύ τολμηρή και προώθησε όσο περισσότερο μπορούσε το θέμα αυτό ώστε να προχωρήσει και έκανε και συγκεκριμένες προτάσεις για το μηχανισμό εγκαίρης προειδοποίησης, αλλά δυστυχώς αυτό δεν φτάνει όσο μακριά θα επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν αποτελεί στην πράξη ένα μηχανισμό αλληλεγγύης. Ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης δεν είναι μηχανισμός αλληλεγγύης και το Κοινοβούλιο εμένει στο γεγονός ότι χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό αλληλεγγύης. Η πραγματική αλληλεγγύη υπάρχει όταν η εισρωή μεταναστών και ετούντων άσυλο είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει ένα κράτος μέλος και υπάρχει βοήθεια. Πριν από μερικές ημέρες υπήρχε μια την αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας ε, στη Λαμπεντούσα και είδαμε ότι η Λαμπεντούσα είναι κενή, διότι παρά το γεγονός ότι 55.000 άνθρωποι ε, κατέφτασαν στις αχθές αυτού του μικροσκοπικού νησιού, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μοιράστηκαν στις διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Οι άνθρωποι όμως που έφτασαν στη Λαμπεντούσα δεν ήθελαν να φτάσουν στη Λαμπεντούσα ούτε καν στην Ιταλία ήθελαν να φτάσουν στην Ευρώπη. Και εάν δεν το κατανοήσουμε, αν δεν αντιληφθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη, θα εξακολουθήσουμε να αφήνουμε τα κράτη-μέλη που βρίσκονται στα σύνορα ε, έρμεα της αντιμετώπισης ε, ε, της εισρωής μεταναστών. Και δεν είναι σωστό αυτό, διότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και η ευθύνη είναι κοινή. Δεν νομίζω ότι ζητά κάποιος από την Ευρώπη να διαιρέσει το οτιδήποτε μεταξύ των κρατών μελών, τον οποιονδήποτε που έρχεται σε ένα κράτος μέλος. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ε, αλληλεγγύης, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν η εισρωή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν μπορεί ένα κράτος μέλος να αντιμετωπίσει τα κύματα μεταναστών μόνο του. Εάν δεν γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να συζητήσουμε πακέτο ασύλου και να συμφωνήσουμε επ' αυτού. Δεύτερον, για τις νέες προτάσεις για τη Σέγγεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε τολμηρές προτάσεις για τη Σέγγεν και η αντίδραση του Συμβουλίου φαίνεται ότι είναι ότι εμείς δεν σα ζητήσαμε να φτάσετε μέχρι αυτού του σημείου. Νομίζω ότι αυτή η αντίδραση από πλευρά Συμβουλίου ήταν απογοητευτική σε κάποιο βαθμό και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε πιο επικοδομητική συνεργασία των νέων ε, σε θέματα αυτές προτάσεων και ε, να συζητήσουμε και το θέμα της εισαγωγής εσωτερικών συνόρων μεταξύ ενός κράτους και άλλου. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι σε αυτές τις προτάσεις για τον απλό λόγο ότι η ελευθερία κυκλοφορίας είναι ένα δικαίωμα το οποίο μας έχει δοθεί σε όλους τους πολίτες μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν θα πρέπει ποτέ να αφαιρέσει κάποιος αυτό το δικαίωμα από μονομερή κίνηση ενός κράτος μέλος. Όταν η Γαλλία ξεκίνησε και εκ νέου τους συνοριακούς ελέγχους με την Ιταλία στις αρχές του έτους, όχι μόνο παραβίαζαν τα δικαιώματα των πολιτών, δικαιώματα τα οποία τους έχει εκχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, αλλά δυστυχώς απέστειλε και ένα πάρα πολύ αρνητικό μήνυμα, διότι μετά από τη Γαλλία είχαμε και τη Δανία και την περασμένη εβδομάδα τις κάτω χώρες. Και το αρνητικό μήνυμα ε, καταδεικνύει ότι αντί να προχωράμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, δυστυχώς έχουμε αρχίσει να οπισθοχωρούμε. Τέλος, για την ε, διεύρυνση και το θέμα του Σέγγεν ζήτησα από την Προεδρία να συνεχίσει το δύσκολο έργο που ανέλαβε και εκτιμώ το γεγονό ότι ήταν πολύ επικοδομητική η προσέγγιση τη, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα έχουν ε, ίσα δικαιώματα στη διεύρυνση ε, της περιοχής Σέγγεν. Ζητάμε από τις χώρες αυτές να δεχτούν και να τηρήσουν προϋποθέσεις και το έκανε. Ελέγξαμε κατά πόσον τήρησαν τις υποχρεώσεις τους και διαπιστώσαμε ότι τις τήρησαν. Τι περιμένουμε λοιπόν, γιατί δεν γίνεται διεύρυνση στην περιοχή Σέγγεν και στις χώρες αυτές, γιατί ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να ε, μπλοκάρει τη διαδικασία όταν οι χώρες αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις. Νομίζω ότι και μόνο για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνει διεύρυνση ε, στις χώρες αυτές, στην περιοχή Σέγγεν, το συντομότερο δυνατόν. Η κυρία Ρωμέρο Λόπεθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να μιλήσω για το σύστημα ασύλου και να επιβεβαιώσω το σχόλιο που μόλις έκανε ο κύριος Μπουσούτιλ. Για τις ελλείψεις που μπορεί να έχει ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης, διότι κατανοούμε μεν τι προσπάθειες έκανε η Πολωνική Προεδρία, αλλά το πρόβλημα έγκυται στον κανονισμό του Δουβλίνου και πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει επιληθεί στο έγγραφο που μας παρουσίασε η Επίτροπος Μάλστρομ αναφέρεται ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου πρέπει να τροποποιηθεί, αλλά δεν μας εξηγεί προς ποια κατεύθυνση. Γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δεν γνωρίζουν τι ακριβώς να κάνουν με τον κανονισμό του Δουβλίνου. Θέλουν να συνεχίσουν να μένει όπως είναι η κατάσταση, δηλαδή οι χώρες του Νότου που ε, δέχονται επίθεση από όλες τις πλευρές της γης, από ανθρώπους που ζητούν άσυλο ε, και έχουν πρόσφυγες και θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να τα αντιμετωπίσουν. Επειδή ακριβώς δεν ισχύουν σωστά τα πράγματα, γίνεται αυτό το οποίο συμβαίνει επί παραδείγματι στην Ελλάδα, στη Μάλτα ή στην Ιταλία, στις χώρες του Νότου που υποδέχονται τόσους πολλούς ε, μετανάστες και δεν έχουν τρόπο να διοχετεύσουν κάπου τα προβλήματά τους. Ε, δεν θα σταματήσει αυτή η διαδικασία εάν ε, δεν κάνουμε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπουσούτιλ να αντιμετωπίσουμε το θέμα ως θέμα λιλεγγύης. Και δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα ρυθμίσουμε με το μηχανισμό εγκαίρης προειδοποίησης. Κατανοούμε την προσπάθεια που έκανε η Πολωνική Προεδρία για το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα το θέμα του ελέγχου των συνόρων, τον εσωτερικό έλεγχο των συνόρων, τον οποίο αναφέρουμε και στην πρόταση οδηγίας που έγινε, και αναφέρθηκε και ο κύριος Μπουσούτιλ στην κατάσταση στη Λαμπεντούζα, είναι αλήθεια ότι δεν μπορεί κάποιο να παρακολύσει την κυκλοφορία προσώπων, αλλά λαμβάνοντα υπόψη και αυτό ω προπόθεση, πιστεύω ότι η Πολωνική Προεδρία έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να μην προχωρήσει η πρόθεση δύο κρατών μελών που αντιμετώπισαν το πρόβλημα και δεν ήξεραν πώς να το επιλύσουν και να αντιληφθούν ότι είναι πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα. Δεν είναι απλώς και μόνο ένα σύνορο, έλεγχος σύνορων. Αναφέρεται και στην οδηγία. Είναι έλεγχος της μετανάστευσης. Μετά βέβαια αναφερόμαστε σε αθλητικές εκδηλώσεις, σε τρομοκρατία και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να, να μιχνιούμε τα πάντα στο ίδιο καζάνι. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα όπως του αρμόζει είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι είναι και θα πρέπει ε, να αποσυρθεί αυτή η οδηγία διότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα με τόσο βεβαιασμένο τρόπο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να παρακολύσουμε την κυκλοφορία των ανθρώπων και από εκεί και πέρα να επεξεργαστούμε αυτό. Όσον αφορά τα στοιχεία PNR, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αναφέρεστε στη διαφάνεια. Πρόκειται για μια διαφάνεια η οποία θα αφορά κυρίως τους επιβάτες, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι θα χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθεσία ούτε καν στο Ηνωμένο Βασίλειο για το PNR η νομοθεσία που αναφέρεται στο Μητρό Επιβατών είναι νομοθεσία τριών ή τεσσάρων χωρών και δεν αφορούν συγκεκριμένα το θέμα των PNR. Υπάρχουν θέματα που αφορούν και τη μετανάστευση και άλλα. Και όσον αφορά ε, τη μετανάστευση, είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση σε αυτές τις τρεις-τέσσερις χώρες. Ε, σε κάποιες είναι για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι για την αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά της ε, δημόσιας τάξεως και σε άλλη περίπτωση περίπτωση είναι το θέμα της μετανάστευσης. Πώς θα έχουμε ευρωπαϊκή οδηγία για το θέμα αυτό όταν δεν υπάρχουν ούτε καν ελάχιστες προδιαγραφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προχωρήσει και θα περάσει πέρα από όλες τις ε, ευρωπαϊκές νομοθεσίες που δεν υπάρχουν και μάλιστα με τελείως διαφορετικά πεδία εφαρμογής. Τι θέση έχει η Πολωνική Προεδρία ή τι θέση ε, κράτησε η Πολωνική Προεδρία για το θέμα αυτό. Η κυρία Βίκστρομ. Ευχαριστώ, Θα μιλήσω σου ειδικά γιατί έχουμε πολύ καλούς διερμηνείς, λέει ευγενικά η ομιλήτρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πολωνική Προεδρία για μια εξαιρετικά αγαστή συνεργασία και για έναν επικοδομητικό διάλογο και για τη διαφάνεια που επικράτησε στις εργασίες της. Αυτή η πνοή διαφάνειας θέλουμε να χαρακτηρίζει το έργο όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και να χαρακτηρίζει όλες τις ε, διαθεσμικές σχέσεις. Ξέρετε, η κρίση που βιώνουμε είναι πολύ περισσότερο από μια οικονομική κρίση. Είναι κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Λυπάμαι και πονάω όταν διαπιστώνω ότι είναι κενή νοήματος ε, η λέξη αλληλεγγύη πλέον. Έχει χάσει, έχει εκφυλιστεί, έχει χάσει την αρχική της έννοια πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αξιοπιστία θα πρέπει να δρούμε με αξιόπιστο τρόπο. Αυτή είναι η λύση. Όμως το αντίθετο επικρατεί σήμερα σε όλα τα κράτη-μέλη. Αναξιοπιστία και έλλειψη εμπιστοσύνης. Ε, και αυτό προκύπτει και από τα πορίσματα πολλών συμβουλίων. Για να ενισχύσουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη ε, των ε, πολιτών θα πρέπει να δράσουμε και αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Ε, όλα αυτά τα υπέροχα λόγια για την αλληλεγγύη δεν μπορούν να μας ικανοποιήσουν γιατί ξέρουμε ότι αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Αυτό το πακέτο με τα πέντε νομοθετήματα σχετίζεται ακριβώς με αυτό το θέμα, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης της πίστης των πολιτών. Μόνο έτσι θα ενισχύσουμε την αλληλεγγύη αυτό που όλοι ε, λένε ότι επιθυμούν. Πολύ σπάνια όμως ε, μιλάμε για αυτές τις ε, σημασιολογικά φορτισμένες λέξεις όπως η αλληλεγγύη μα είναι ε, θέμα ανθρωπιάς. Ξέρετε ότι οι άνθρωποι που έρχονται στην Ήπειρό μας αυτό αποζητούν να αισθάνονται σιγουριά και να έχουν εμπιστοσύνη στους ηθήνοντες. Εγώ είμαι υπεύθυνη για τον κανονισμό Δουβλίνου. Χαίρομαι για τα αποτελέσματα των εργασιών του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι για τη συνεργασία που είχαμε, χάρη στην οποία Σύντομα μπορούμε να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του κανονισμού. Λοιπόν, θα ήθελα να δράξω τη σημερινή ευκαιρία και να τονίσω ότι για την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξουμε φρασιολογίες που τονίζουν ακριβώς αυτό που σας είπα, δηλαδή ενισχυμένη αλληλεγγύη που βασίζεται σε ενισχυμένη πίστη ε, ε, από πλευράς ε, των πολιτών. Εμπιστοσύνη. Και γι' αυτό θα πρέπει να χωρίσουμε την συζήτηση για τον κανονισμό ε, του Δουβλίνου από όλα τα υπόλοιπα νομοθετήματα. Θα πρέπει ξεχωριστά να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον, ε, τους εισηγητές και τους σκιώδης εισηγητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Επίσης σημαντικό ήταν το έργο της Πολωνικής Προεδρίας για την Ένωση και ευχαριστώ τον Υπουργό για την διεξοδική παρουσίαση που έκανε για όλα τα επιτεύγματα του τελευταίου εξαμήνου στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνη. Είναι καθοριστική σημασία αυτά τα ζητήματα για το μέλλον μα. Ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια για του πολίτε τη Ένωση είναι ζήτημα προτεραιότητα για μα. Δεν έχουμε όμω ολοκληρώσει τι προσπάθειέ μα, ούτε έχει ολοκληρώσει η Προεδρία σα. Στι 30 Δεκεμβρίου, λοιπόν, στο Συμβούλιο, ε, σας καλώ να μιλήσετε ακριβώς για αυτό το θέμα, για το πώς θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών για να εκλείψει αυτή η έλλειψη πίστης που χαρακτηρίζει τους πολίτες, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και να κινηθούμε όλοι από κοινού που να κατανοήσουν τα κράτη-μέλη ότι ε, εν τη ισχύ δύναμη δεν γίνεται να προχωρήσουν, ενώ ή δύναμη, ήθελα να πω, ζητώ συγγνώμη, δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν μόνα τους και προς αυτό θα πρέπει να αποσκοπούν τα νέα ε, νομοθετήματα. Θα ήθελα λοιπόν στον υπόλοιπο χρόνο της Προεδρίας σας, έστω και να αυτός είναι περιορισμένος, για το πακέτο ασύλου και για την έκθεση για την οποία είμαι αρμόδια να μεριμνήσουμε όλοι μαζί ώστε να επικρατήσει αυτή η πνοή ε, εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης ε, και διαφάνεια στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε κυρία Βίξτρομ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις... Θα δώσουμε τις απαντήσεις. Ένας πρώτος γύρος απαντήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχήν να απαντήσω στις ερωτήσεις που έγιναν με τη σειρά που έγιναν, ξεκινώντας με ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά είναι εμφανές σε όλες τις ερωτήσεις το θέμα του Δουβλίνου. Συνειδητοποιώ ότι όλες οι προσδοκίες για αλλαγή, για τροποποίηση αυτής της νομοθεσίας, αυτών των κανονισμών, δεν έχουν ικανοποιηθεί. Εμείς κάνουμε μια σαφή αναφορά στο θέμα αυτό στα εισαγωγικά μας σχόλια, θεωρώντας ότι πρόκειται για τη βάση των αλλαγών που έγιναν. Παρ' όλα αυτά, αναφερθήκαμε και στην καρδιά του εγγράφου και όχι μόνο στην εισαγωγή, όπου υπάρχει η πρόταση για ένα άρθρο που αφορά πολύ συγκεκριμένα τους μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης, αλληλεγγύης και άλλες τροποποιήσεις και τροπολογίες, οι οποίες όμως, αν θέλετε, δεν έχουν προχωρήσει καθότι η τροποποίηση αυτού του άρθρου έχει σταματήσει. Κατά τη διάρκεια του επόμενου Συμβουλίου πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί και ενδεχομένως θα προετοιμαστεί μια νέα σύνταξη του κειμένου, του άρθρου, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα αυτό. Βεβαίως η αλληλεγγύη στην Ευρώπη δεν περιορίζεται και δεν σταματά σε καμία περίπτωση στο Δουβλίνο. Χρειάζονται και άλλα κείμενα τα οποία θα πρέπει να προετοιμαστούν τα επόμενα χρόνια. Την Παρασκευή Εξάλλου είδαμε και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το άσυλο και την αλληλεγγύη. Υπάρχει σειρά κειμένων και προτάσεων που αντικατοπτρίζουν τα θέματα αυτά, θέματα που αφορούν την αλληλεγγύη, την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και θέματα διακυβέρνησης ε, που αφορούν το Σέγγεν. Ο Ντόναλτ Τούσκ έχει αναφερθεί πολύ πρόσφατα στο θέμα αυτό. Η πολωνική θέση είναι σαφής. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη επεξεργάστηκαν τα κείμενα και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πολύ μεγάλη προσοχή και επιφύλαξη όσον αφορά τους μηχανισμούς που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και ιδιαίτερα σε περίπτωση παράνομης μετανάστευσης. Και βεβαίως εδώ η μηχανισμοί και η αντιμετώπιση θα πρέπει να είναι κοινοτική και όχι εθνική η αντιμετώπιση. Το θέμα είναι πώς να οργανωθεί κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι μετά την συνάντηση κορυφής της επόμενης εβδομάδας περιμένουμε και προσδοκούμε να υπάρξει ένας οδικός χάρτης, ένας χάρτης πορείας, βάσει του οποίου θα συνεχίσουμε την εργασία μας στον τομέα αυτό. Και βεβαίως η Πολωνική Προεδρία έχει προχωρήσει πολύ προσεκτικά στην επεξεργασία αυτών των θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς αυτό που είπατε. Δεν υπάρχουν λύσεις στα κράτη-μέλη μεμονωμένα. Ακούσαμε κάποιες θέσεις, υπήρξαν φυσικά διαβουλεύσεις με τους χρήστες, με τις αεροπορικές εταιρείες για θέματα PNR και βεβαίως όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες εργασίας και σε αυτές τις διαβουλεύσεις, όλα τα συμβαλόμενα μέρη υπέβαλαν τις προτάσεις τους και η βάση στην οποία μπορούμε να εργαστούμε από εδώ και πέρα είναι το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας. Αυτή η εργασία πρέπει να σας πω έγινε πολύ προσεκτικά, πολύ αργά, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα θέματα. Η διεύρυνση του Σέγγεν. Άλλο θέμα. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε προβλήματα στον τομέα αυτό. Η Προεδρία έκανε ό,τι μπορούσε υποβάλαμε συμβιβαστικές ε, λύσεις. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία βεβαίως δεν μπόρεσαν να δεχτούν αυτή τη συμβαστική λύση. Περίμεναν κάτι τελείως διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να συμφωνήσουμε με τις χώρες αυτές, με τις χώρες που δεν ήθελαν να διευρυνθεί το Σέγγεν από την άλλη μεριά. Επίσης μπορέσαμε να βρούμε μια συμβαστική λύση. Από την άλλη μεριά η συνθήκη είναι σαφής. Χρειάζεται εδώ ομοφωνία. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε ομοφωνία. Προς το παρόν τουλάχιστον και κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής του Σεπτεμβρίου ομοφωνία δεν επετεύχθη. Συνεχίσαμε λοιπόν τις συζητήσεις, τις διαβουλεύσεις από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα και ελπίζω σε ένα υψηλότερο επίπεδο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων θα μπορέσουν να υπάρξουν πραγματικά σημαντικές αλλαγές. Από ό,τι ξέρω, το θέμα αυτό θα είναι στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Συμβουλίου. Η νομοθεσία σήμερα πάντως παρόλες τις προσπάθειες της πολιτικής Προεδρίας δεν έχει αλλάξει, δεν έχει τροποποιηθεί. Η ημερήσια διάταξη, αν θέλετε, της Πολωνικής Προεδρίας μέχρι τα Χριστούγεννα συμπεριλαμβάνει περισσότερες προσπάθειες και δεν πρόκειται να σταματήσουμε μέχρι την τελευταία ώρα της Προεδρίας μας αυτές τις προσπάθειες. Κατά την άποψή μας μπορέσαμε να δημιουργήσουμε εξαιρετικές σχέσεις εργασίας, συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνεχείς επαφές και μια πραγματική συνεργασία που μας επέταξε, που μας ε, βοήθησε να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο σε πάρα πολλά θέματα και γι' αυτό και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Όχι, ο κύριος Μπουσούτιλ. Επιτρέψτε μου να κάνω μία έκκληση προς την Προεδρία. Ήσασταν πάντα επικοδομητικός, ανοιχτόμυαλος, ε, ε, συγγνώμη, στην Προεδρία. Ήταν, ήταν πάντα επικοδομητική ως Προεδρία και σας προτρέπω να παραμείνετε ακόμα επικοδομητικός και ανοιχτό μυαλός, ακόμα και όταν θα αναλάβετε και πάλι τη θέση σας ως απλό μέλος του Συμβουλίου Υπουργών μετά από τη λήξη της Προεδρίας σας. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, Λέει ο Πρόεδρο, είμαι βέβαιο ότι και οι δύο εκπρόσωποι της Πολωνικής Προεδρία σημείωσαν ότι εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την επικοδομητική του προσπάθεια και το ευρωπαϊκό πνεύμα το οποίο επέδειξαν. Όπως σας είπα προηγουμένως, με το πνεύμα αυτό διεξήγαγαν τα καθήκοντά τους ε, στη διάρκεια αυτού του δύσκολου εξαμήνου, προχωρούσαν ε, τα ακαθόδη ζητήματα και εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι ήταν ειλικρινής και έντιμη προς την Επιτροπή μας ε, όταν συζητούσαμε απτά προβλήματα και προσκόμματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. have not Στη διάρκεια της Προεδρίας δεν παρουσίασαν τις δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν ως κάτι ίσονο σημασία και φυσικά μπορέσαμε έτσι να προχωρήσουμε όλα τα θέματα τα οποία ήταν ουσιαστικά για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στη διάρκεια του εξαμήνου. Αν θέλετε να δώσετε μια τελευταία πινελιά, κύριε Σταχάντση και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ εν είδη συμπεράσματο, θα ήθελα να απαντήσω και σε αυτά που μόλι είπατε και εσεί, κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να σα ε, εγγυηθούμε ότι η Πολωνία θα μείνει ίδια. Θα είναι μια αντιπροσωπεία ε, υπέρ της Ευρώπης και με υποδομητικό πάντα πνεύμα, ανεξάρτητα από το ποιος θα έχει τα ενία στην Προεδρία. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Υπάρχει ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη αλλά έχει προγραμματιστεί για τρι, ε, τις 6 ε, παρατέταρτο. Ο πρέσβης της Βραζιλίας δεν είναι εδώ ακόμα. Ε, τον έχουμε ζητήσει επανειλημμένως να παραστεί για να συζητήσουμε θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και δεν έχει έρθει ακόμα. Προτείνω λοιπόν να κάνουμε ένα διάλειμμα για τρία τέταρτα Μισή ώρα. Για 20 λεπτά. Διακόπτουμε λοιπόν για 20 λεπτά. Έχετε αρκετό χρόνο να ασχοληθείτε με άλλα θέματα λοιπόν. Σας παρακαλώ όμως να είστε πίσω σε 20 λεπτά, διότι θα γίνει και συνεδρίαση συντονιστών αμέσως μετά την παρουσία του πρέσβη. Ευχαριστώ πολύ.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 the minister in the attendance to this part of the... Έχουμε λίγους ε, παρισταμένους σε αυτό το τμήμα της συνεδρίασης. Καλωσορίζουμε παρόλα αυτά τον κύριο Νέιβα Ταβάρες, πρέσβη της Βραζιλίας, ο οποίος ε, προσεκλήθη να συμμετάσχει στην σημερινή συνεδρίαση για μια ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα αμοιβαιότητα στην πολιτική θεωρήσεων ασφάλειας, τρομοκρατίας και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο κύριος Ρικάρντο Νέιβα Ταβάρες είναι πρέσβης της Βραζιλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε λάβει την πρόσκλησή μας ε, για να μπορέσει να συζητήσει θέματα τα οποία έχουμε στην ημερήσια διάταξη εδώ. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα διότι βρήκε το χρόνο να έρθει. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας, η οποία έγινε στις 4 Οκτωβρίου, και οι δύο πλευρές, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βραζιλία, επιβεβαίωσαν εκ νέου την διάθεσή τους να συζητήσουν ε, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και εγκάρσεων προκλήσεων όπως για παράδειγμα η διαφθορά, η νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων και η, το εμπόριο ναρκωτικών. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον πρέσβη και κατόπιν θα ξεκινήσει ένας γύρος ε, παρεμβάσεων για τα μέλη που θέλουν να παρέμβουν. Παρακαλώ κύριε πρέσβη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ενημερώθηκα ότι μπορώ να μιλήσω πορτογαλικά. Τέλος πάντων, βραζιλιάνικα, πορτογαλικά θα μιλήσω. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω σήμερα στις εργασίες της Επιτροπής σας, τα θέματα αρμοδιότητά σας, δηλαδή ότι άπτεται του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, συνιστά και την πεμπτουσία της ε, στρατηγικής εταιρικής σχέσης ε, ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση μας βασίζεται στη συγγένεια των αξιών και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ιστορία της Βραζιλίας χαρακτηρίζεται από τη διαρκή αναζήτηση μιας πιο αποτελεσματικής άσκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε αυτόν τον αγώνα συμμετείχε προσωπικά η πρόεδρος της Δημοκρατίας Ντίλμα Ρουσέφ, όπως σίγουρα γνωρίζουμε τα μέλη της Επιτροπής σας. Ο επανεκδημοκρατισμός της χώρας από τα μέσα τη δεκαετία του 80 και μέχρι σήμερα δεν θα είχε ολοκληρωθεί αν εξακολουθούσαν να υπάρχουν αυτά τα ανησυχητικά επίπεδα κοινωνική ανισότητα. Για την ε, Βραζιλία δεν υπάρχει καμία ιεράρχηση ανάμεσα στα πολιτικά δικαιώματα αφενό και τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα αφετέρου. Στη δεκαετία των 90 κατοχυρώσαμε την νομισματική σταθερότητα και με υψηλά αναπτυξιακά ποσοστά τελικά η χώρα μας μπόρεσε να ασχοληθεί με τη μείωση της ευτόχειας και της έλλειψης δικαιοσύνης. Από το 2003 μέχρι το 2010 20 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι ξέφυγαν από την ε, ακραία φτώχεια και περίπου 40 ε, εκατομμύρια εισήλθαν στη μεσαία τάξη, η οποία τώρα αντιστοιχεί στο ίμιση του πληθυσμού της Βραζιλίας. Έχουμε κοινέ αρχές, όπως έλεγα προηγουμένως, που σχετίζονται σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ε, πολυμερή φόρα. Έχουν ήδη συνεδριάσει τρει φορέ οι εμπειρογνώμονε και από τι δύο πλευρέ ε, στα πλαίσια του διμερούς ε, τομεακού διάλογου, διαλόγου συγγνώμη, το 2008. Από πλευρά μα εκπροσωπήθηκε η Βραζιλία από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον πρέσβη δηλαδή Αντώνιο Πατριώτα και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχαμε την ύπατη εκπρόσωπο Κάθριν Άστον και συζητήσαμε τα θέματα ε, κοινού ενδιαφέροντο. Η Βραζιλία δηλώνει αλληλέγγυα ε, προς όλες τις χώρες ε, που διεκδικούν τη δικαιοσύνη και την ε, ελευθερία τους. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται στην άσκηση βίας και στην καταστολή. Καμία ηγεσία δεν μπορεί να βασιστεί στην κοινωνική αποξένωση, στην ανεργία και στην φτώχεια. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε καμία περίπτωση σε παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων των πολιτών μας. Επανειλημμένα η κυβέρνηση της Βραζιλίας έχει συμμετάσχει σε δράσεις αλληλεγγύη και σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης υπέρ της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην ε, Βόρεια Αφρική και στην ε, Μέση Ανατολή σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί μας ούτως ώστε να προβούμε στις ε, απαιτούμενες ε, μεταρρυθμίσεις, χωρίς να ξεχνάμε όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται επιβολή άδικων κυρώσεων, ούτε στρατιωτική επέμβαση. Όπως είπε η πρόεδρος Ντίλμα Ρούσεφ ε, το Σεπτέμβρη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και παραθέτω, υποφέρει ο κόσμος από τις επώδυνες επιπτώσεις των στρατιωτικών παρεμβάσεων που κλιμάκωσαν τις διενέξεις, επέτρεψαν τη, να διεισδύσει στις χώρες ο, η τρομοκρατία, συγγνώμη, και να άρχισαν νέους κύκλους βίας. τέλο παράθεση. Χρειαζόμαστε λοιπόν διπλωματικά και ανθρωπιστικά μέσα για να δράσουμε. Μόνο όταν δεν επαρκούν τα ειρηνικά μέσα, μόνο σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο χρήση κατασταλτικών μέτρων ε, για να ε, ε, προστατεύσουμε τη συλλογική ασφάλεια, όπως προτείνει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε φυσικά την ευθύνη να προστατεύσουμε τους ε, πολίτες, αλλά μην ξεχνάμε και την ε, ευθύνη ε, που έχουμε κατά τη διάρκεια της προστασίας. Δηλαδή όταν κρίνεται απαραίτητη η άσκηση της βίας θα πρέπει να την ελαχιστοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού. Ε, που δεν είπε η στρατιωτική παρέμβαση δεν πρέπει να προκαλέσει μεγαλύτερα δεινά από αυτά που αρχικά είχε ως στόχο να καταπολεμήσει. Λοιπόν η συλλογική δράση πρέπει να είναι αποτελεσματική, αναλογική και περιορισμένη στους στόχους όπου και ορίζει το Συμβούλιο, της, ε, Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρέπει να θυμόμαστε επίση ότι η κοινωνική αποξένωση σπάνια συνοδεύεται από σταθερότητα και από ασφάλεια. Δίκιο έχει ο Γενικό Γραμματέας του ΟΗΕ που λέει και παραθέτω η ανάπτυξη είναι καλύτερη πρόληψη. Κλείνω την παράθεση. Άλλα μέσα επίση είναι στη διάθεση τη διεθνού κοινότητα, Παραδείγματο χάρη ειρηνευτικέ διαδικασίε που απέδειξαν την αξία του ω ε, ε, αποτελεσματικά μέσα σε πολλέ περιπτώσει. Μην ξεχνάμε όμω και τον αφοπλισμό και την καταστροφή ε, των όπλων μαζική καταστροφή που επίση μπορεί να συμβάλλουν το μάλλον στη διατήρηση ειρήνης. Ε, η Βραζιλία ε, καταδικάζει απερίφραστα την άσκηση της βίας. Αυτό καταδικάζει τούτο ή άλλως από το Σύνταγμά μας και χαρακτηρίζει όλε τι διεθνείς σχέσει μα Έχουμε προσχωρήσει σε όλε τι συμβάσει συμβάσεις τα διεθνή πρωτόκολλα που σχετίζονται με την απειλή της βίας. Το φάσμα τη τρομοκρατίας επίση αποτελεί για ρήξη και μορφέ συντονισμού τη δράση ανάμεσα στα κράτη. Εμείς υποστηρίζουμε την παγκόσμια στρατηγική κατά της τρομοκρατίας ε, του ΟΗΕ που στόχο έχει να ενισχύσει τις, ε, τα εθνικά μέσα πρόληψης αλλά και να ε, μεριμνήσει ώστε να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να επικυρωθεί μια ευρεία εφαρμογή σύμβαση του ΟΗΕ κατά τη, του, της διεθνούς Επίσης, άλλα θέματα που μας απασχολούν είναι η χρηματοδότηση χρηματοδότηση της τρομοκρατικής δράσης και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και το, η Βραζιλία ανήκει στο FATF, ε, που είναι η διεθνή Ομάδα χρηματοπιστωτική δράση, που στόχο έχει την πρόθεση των πολιτικών για την καταπολέμηση του ξέπλυματος ε, βρώμικου χρήματο και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Επίση ανήκουμε στην FATF ε, Sud, δηλαδή όπου συμμετέχουν όλε οι χώρε τη Λατινική Αμερική, έχοντα του ίδιου στόχους. Ε, συμμετέχουμε επίση ε, και στην ομάδα Egmont ε, με υπηρεσίε πληροφοριών σε χρηματοπιστωτικά θέματα από δεκάδε χώρε. Το η Βραζιλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, και την τήρηση του διεθνούς ε, δικαίου ε, και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι αλληλοσυμπληρούμενοι αυτοί οι στόχοι, διότι ναι, πρέπει να καταπολέσουμε την τρομοκρατία, αλλά θα πρέπει να θέτουμε την, τον αγώνα αυτό κατά της τρομοκρατίας στην πολιτική ηγεσία και να διατηρούμε ταυτόχρονα την τάξη. Ε, συμπίπτουν λοιπόν τα οράματα τη Βραζιλίας και τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω προ την διμερή συνεργασία για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Μην ξεχνάτε ότι στην ιστορία μας υπάρχουν ε, εκατομμύρια μάρτυρε, δηλαδή ε, μετανάστες ε, που έχουν έρθει από όλες τι γωνιέ του κόσμου, προσπάθησαν να βρουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και με την δουλειά, την έντιμη δουλειά του μπόρεσαν να ενσωματωθούν στην κοινωνία τη Βραζιλία. Μην ξεχνάτε ότι η πρόεδρο μα, καθώ και ο αντιπρόεδρο Μισελ Τέμερε είναι βραζιλιάνη πρώτης γενιάς. Έτσι φαίνεται πόσο ανοιχτή είναι η κοινωνία της Βραζίλία, Ο, ο πατέρας της κυρίας Ρουσέφ, παραδείγματος χάρη, ήταν δικηγόρο στη Βουλγαρία και έφυγε από την Ευρώπη διότι έψαχνε μια καλύτερη ζωή στη Λατινική Αμερική. Από τις αρχές του, ε, της δεκαετίας του 80 έχουν σημειωθεί πολλές αλλαγές ε, και στις αρχές της δεκαετίας του 80 υπήρχαν περισσότεροι Βραζιλιάνοι μετανάστες ε, που έφευγαν από τη χώρα από ότι οι μετανάστες που έφταναν στη Βραζιλία. Ελπίζουμε λοιπόν ε, να τύχουν υποδοχή σε αυτοί οι μετανάστες στις άλλες χώρες, ε, όπως ε, επιφυλάξαμε και εμείς σε πολύ καλή υποδοχή σε όλε τι μετανάστες που κατέφυγαν στην Βραζιλία. Τώρα έχουν ανατραπεί οι τάσει, και τώρα και πάλι ο αριθμός των Βραζιλιάνων που φεύγουν από τη χώρα είναι χαμηλότερος από τον αριθμό αυτό των μεταναστών. Το μεταναστευτικό φαινόμενο όμως είναι ευμετάβλετο, έχει μια δική του δυναμική και η Βραζιλία θεωρεί ότι στον τομέα της μετανάστευσης και πέραν κάθε άλλης ανησυχίας θα πρέπει να φροντίζουμε να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και των οικογενειών τους ανεξαρτήτως εθνικότητας, ε, κατάστασης, εθνικής ενωτικής προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Μας ανησυχούν όμως οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ποινικοποίηση της παράνομης μετανάστευσης. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα παραδείγματος χάρη σε κάποιον που δεν έχει ε, ε, νόμιμη διαμονή σε μια χώρα και κάποιον ε, που εμπλέκεται σε εγκληματικές δραστηριότητες. Μπορεί κάποιο να μην έχει τα πετούμενα έγγραφα αλλά να εργάζεται έντιμα και προ... υπάρχει μεγάλη διαφορά λοιπόν ανάμεσα σε αυτόν και σε κάποιον που εμπλέκεται σε παράνομες και διεγκληματικές δραστηριότητες. Η εργαστές ε, συμμετέχουν στην κοινωνία υποδοχής ε, χάρη στη δουλειά τους, ε, το δυναμισμό τους και την πολιτιστική τους κληρονομιά ε, παρόλα αυτά βρίσκονται σε μια επισφαλή θέση και εκτίθενται ε, σε αδίστακτους ε, εγκληματίες ε, και γνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα ήδη έχουμε εφαρμόσει τα προγράμματα νομιμοποίησης. Το 2009 παραδειγμα χάρη νομιμοποιήσαμε πάνω από 41.000, 41.800 αλλοδαπούς. Θέλουμε να ενισχύσουμε επίσης την αστυνομική συνεργασία για την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων διακίνησης μεταναστών. Θα θέλαμε λοιπόν σε διμερέ και πολυτιμερέ επίπεδο να συνεχιστεί η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευση ε, και να προστατεύσουμε αυτούς του μετανάστες ανεξαρτήτως ε, εθνικότητας. Ε, δεν μπορούμε επίση να επεμβαίνουμε στις προσωπικές αποφάσεις ε, των πολιτών μας. Οι Βραζιλιάνοι μπορούν να ταξιδεύσουν και να διαμείνουν σε οποιαδήποτε χώρα θέλουν. Ε, δεν μπορούν οι δημόσιε αρχέ να του περιορίσουν οδήποτε τρόπο. Φυσικά, η κυβέρνηση τη Βραζιλία μπορεί να ενημερώσει τους ταξιδιώτε σχετικά με τις συνθήκες εισόδου στις χώρες. Έχουμε ήδη οργανώσει σεμινάρια σε διάφορε πόλει όπου διαπιστώθηκε ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στρέφεται και φεύγει σε ξένε χώρες. Όμως ε, το Υπουργείο Εξωτερικών πρόσφατα εξέδωσε ε, το εγχειρίδιο επανόδου στη Βραζιλία ούτως ώστε να ε, υποδεχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτούς που επιστρέφουν στη χώρα. Επίσης, θα να σχολιάσω τη διμερείς συμφωνίας για τις σύντομες διαμονές που έχει υπογράψει η Βραζιλία με 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε ε, ε, κλείσει τι συμφωνίε με τέσσερι χώρες, η Κύπρο, Εσθονία, ε, Λιθουανία και Μάλτα και τελικά όμως λόγω της εφαρμογής ε, του κοινοτικού και εκτιμένου και μετά την προσχώρηση αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώθηκαν συμφωνίες και με αυτές τις χώρες. Ε, θα θέλαμε επίσης να ενταχθούν, ε, να αντικατασταθούν μάλλον αυτές οι διμερείς συμφωνίες από μια διεθνή συμφωνία, διότι δημιουργείται μια κατάσταση να, μη συγγνώμη αμοιβαιότητας που δεν έχει προκαλέσει η Βραζιλία. Οι αρχές της Βραζιλίας λοιπόν και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν αρχίσει ήδη τις ε, για την συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ε, και τελικά έχουν υπογραφεί και εφαρμόζονται σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία με τις οποίες, για τις οποίες ισχύουν ακόμη οι διμερείς, οι πρώτερες διμερείς συμφωνίες. Οι νέες συμφωνίες ε, φυσικά δεν αλλάζουν σε τίποτα την κατάσταση των επισκεπτών προέρχονται από την Βραζιλία, ούτε αλλάζουν τίποτα για τους αυτών των 23 ε, κράτων που έχουν προσυπογράψει τις ευημερείς ε, αυτές ε, συμφωνίες. Επίσης, σε αυτό το νέο μηχανισμό διευκόλυνσης του ταξιδιού συμπεριλαμβάνονται οι υπήκοοι και αυτών των τέσσερων κρατών και υπενθυμίζω ότι μας συνδέουν σχέσεις φιλίας με αυτές τις τέσσερις χώρες. Υπεγράφησαν τον περασμένο Νοέμβριο αυτές οι συμφωνίες. Χαιρόμαστε και ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την τοποθέτησή του, διότι έδωσε τη σύμφωνη γνώση η Επιτροπή σας για την υπογραφή αυτών των συμφωνιών. Πρόκειται για δύο διαφορετικές Ευρωπαϊκή Συμφωνία σε μία για τα διπλωματικά επίσημα και υπηρεσιακά διαβατήρια που ισχύει ήδη από τον Απρίλιο το 2011 και μία άλλη συμφωνία για τα, ε, διαβατήρια, τα κοινά διαβατήρια που ακόμη εξετάζεται από την γερουσία μας. Ε, δεν μπορούμε να προδικάσουμε την εξέλιξη αυτής τη διαδικασίας λόγω της ανεξαρτησίας του νομοθετικού, ε, της νομοθετικής εξουσίας. Παρόλα αυτά παρακολουθούμε εκ του σύνεκης και επιθυμούμε μελητή να εφαρμοστούν ε, συγγνώμη, να ε, ε, υπογραφούν αυτές τις συμφωνίες. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να εξετάζει συμφωνίες και σχέσεις όπως αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση που υπάρχει με την Βραζιλία και θα θέλαμε να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Τώρα... Το λόγο έχει ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε την παρουσίαση του πρέσβη που στην πραγματικότητα απλώς ε, παρακολουθήσαμε ε, στα η διάρκεια του έτους διότι επανειλημμένως σας είχαμε ζητήσει να έρθετε εδώ και επιτέλους μας δίνετε αυτή η ευκαιρία. Τη ευκαιρία την οποία θέλουμε να καλλιεργήσουμε μέχρι τέλους. Ακούσαμε τις απόψεις σας για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, για τα σημαντικά βήματα τα οποία καταγράφησαν 40 ε, εκατομμύρια για παράδειγμα άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται πλέον στη μεσαία τάξη. Εγνωρίζουμε πόσο πολύ αναπτύχθηκε οικονομικώς η Βραζιλία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα ε, ως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, αν μου επιτρέπετε και ως ε, Ιταλός πολίτης ο οποίος σήμερα εκπροσωπεί την Ιταλία στην Ευρώπη. Εμείς ε, ακούσαμε την άποψή σας για κάποια ουσιώδη ζητήματα, ε, θεωρήσεις, ε, θέματα ασφάλειας, διαβατήρια και φυσικά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε κάποιες απόψεις από σημαντικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, όπως για παράδειγμα η Justice Global Connectors, η οποία διαπιστώνει όπου υπάρχει μια υποδομή ε, η οποία θα μπορούσε να φιλοξενήσει το πολύ 100 άτομα και στα οποία είχατε συσσωρεύσει 268 άτομα και μάλιστα πρόσχεται για μια φυλακή και θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε κατά πόσον γίνεται κράτηση υπό αυτού τις ώρες. Πώ γίνεται ένα τρομοκράτη ο οποίο έχει καταδικαστεί δι και έχει και ε, καταδικαστική απόφαση από το δικαστήριο μπορεί να βρίσκεται σε τέτοιε φυλακέ οι οποίε έχουν μαζική παρουσία κρατουμένων και όχι ε, σε κάποιο άλλο σοφρονιστικό κατάστημα στο οποίο ε, θα έπρεπε να βρίσκεται στην Ιταλία πιο συγκεκριμένα όπου οι συνθήκες είναι πολύ πολύ πιο αξιοπρεπείς. Επίσης, διαρωτώμεθα πώς γίνεται εσεί σήμερα στην παρέμβασή σας αναφερθήκατε εν γέννη στις ανάγκες συνεργασίας. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα ε, κάποιες πολύ σημαντικές συμφωνίες για θέματα αμοιβαιότητας στις θεωρήσεις. Εσείς μας λέτε ότι δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε την ε, παράνομη μετανάστευση. Ωστόσο, το θέμα αυτό μας οδηγεί σε μια άλλη αξιολόγηση. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που ζουν στη Βραζιλία που είναι Ιταλοί. Πώς είναι δυνατόν ένας τόσο σημαντικός πόρος για τον παραγωγικό ιστό, για την ε, απασχόληση και την ανάπτυξή τους, για τον παραγωγικό ιστό της χώρας, να μην λήφθηκε υπόψη όταν θέλαμε να ε, επιβληθεί μια καταδικαστική απόφαση που ζητούσε την έκδοση του Μπατίστη. Ξέρετε ότι ο Μπατίστη τώρα θα είναι εξαπλωμένος στις παραλίε, έχει γίνει και συγγραφέα. Γνωρίζουμε επίσης ότι ήθελε να επιστρέψει στην Ευρώπη αλλά στη Γαλλία. Γνωρίζουμε δε ότι από ό,τι φαίνεται ο εισαγγελέα ζήτησε να του αρνηθεί το δικαίωμα θεώρησης διαβατηρίου. Αν όντω λοιπόν υπάρχει όπως θα έπρεπε να υπάρχει αμοιβαιότητα και πολύ καλή συνεργασία διότι οι διεθνείς ε, συμφωνίες επιβάλλουν μια συνεργασία που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, σας ρωτώ κύριε Πρέσβη, πώς είναι δυνατόν ακόμα και τώρα για αυτή την υπόθεση Μπατίστη να έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Διότι όταν ε, ε, χάνονται ανθρώπινες ζωές, η δικαιοσύνη πρέπει να ε, πράξει τα δέοντα. Έχουν περάσει 30 χρόνια και ακόμα δεν έχει απονομηθεί η δικαιοσύνη. δε θα θέλαμε λοιπόν να διαποφασίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η οποία δικαστήριο θα επιβεβαιώσει ότι αυτή η αμοιβαιότητα και συνεργασία που ελπίζετε και εσείς και εμείς δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη για μια συνειδητή απόφαση της Βρεοζηλίας, η οποία δεν μας βρέσκει σε καμία περίπτωση σύμφωνος. Ε, κάτι το οποίο βρήκα περίεργο και θα τελειώσω με αυτό κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, ε, κύριε Πρέσβη, υπάρχει θέμα θεωρήσεων και οι Γάλλοι πολίτες έχουν δικαίωμα θεώρησης για 180 μέρες, ενώ κάποιοι άλλοι πολίτες ε, οι Ιταλοί στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν υποβαθμιστεί μετά από αυτή την υπόθεση Μπατίστη και λαμβάνουν μόνο θεώρηση ε, διαβατηρίου για τουριστικούς σκοπούς για 90 μέρες. Ευχαριστώ κύριε Μπουσούτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον πρέσβη που ήρθε τόσο αργά να μας παρουσιάσει αυτά τα θέματα εδώ στην Επιτροπή. Μιλήσατε για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ξέρετε ότι πρόκειται για ένα θέμα μία βεβαιότητα. ιδιαίτερα για τέσσερις χώρες, Εστονία, Λετωνία, Μάλτα και Κύπρος. Η χώρα μου είναι μία από αυτές τις τέσσερις. Αυτό σημαίνει ότι για έναν Βραζιλιάνο μπορεί να επισκεφτεί αυτές τις χώρες χωρίς θεώρηση, χωρίς βίζα, αλλά ότι οι υπήκοοι αυτών των χωρών χρειάζονται βίζα για να επισκεφθούν τη Βραζιλία. Και όντως υπάρχει η συμφωνία η οποία κυρώθηκε από το Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο αυτού του χρόνου. Και από ό,τι ξέρω μέχρι τώρα η συμφωνία αυτή δεν έχει κυρωθεί από την νομοθετική αρχή της Βραζιλίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους ταξιδιώτες οι οποίοι είναι κάτοχοι ενός κανονικού διαβατηρίου και θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα σας. Δηλαδή συνεχίζει αυτή η άδικη κατάσταση, δεν υπάρχει αμοιβαιότητα και το θέμα είναι ότι κάποιοι από τις χώρες μας πιστεύουν ότι πλέον δεν υπάρχει υποχρέωση θεώρησης, μπορεί λοιπόν να ταξιδέψουν, να έρθουν στη Βραζιλία και να τους στείλουν πίσω. Αυτό συνέβη σε κάποιους Μαλτέζους. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, αυτή η συμφωνία γιατί ακόμα δεν έχει κυρωθεί από την νομοθετική αρχή της χώρας σας και πότε θα το κάνετε έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική αμοιβαιότητα όσον αφορά την υποχρέωση θεωρήσεων. Η κυρία Κόνς. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρόμοια ερώτηση με αυτήν του κυρίου Μπούζοτιλ. Αναφερθήκατε στις τέσσερις χώρες και είπατε ότι όσον αφορά τις θεωρήσεις πρέπει να επικρατήσει αμοιβαιότητα. Πότε, για ποιο λόγο, σε τι δυσκολία έχετε πέσει και δεν μπορείτε να επιβάλλετε αυτή την αμοιβαιότητα. Θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα ποιες είναι οι δυσκολίες που σας εμποδίζουν να κυρώσετε αυτή τη συμφωνία. Ο κύριος Ταβάρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, Πρέσβη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω εδώ στην Επιτροπή μας βλέπω να εκπροσωπείται η Βραζιλία στην Επιτροπή. Ε, ξέρετε, χαίρομαι γιατί με συνδέουν πάρα πολλά με την Βραζιλία ως προς την εκπαίδευσή μου, προσωπικές σχέσεις. Ε, τέλος πάντων, έχω οικογένεια, συγγενείς στη Βραζιλία. Ε, Όντω έχει ζήσει μεγάλες αλλαγές η Βροσλία, όχι μόνο οικονομικές ε, και κοινωνικές, ε, αλλά κατοχυρώθηκε πια το κράτος δικαίου, οι πολιτικές ελευθερίες, τα δικαιώματα του πολίτη, παραδείγματος χαρή πολυφωνία στον τύπο, κάτι που συνεχίζεται εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές παρατάξεις από ε, αυτές ε, που τάσσονται υπέρ της κυβέρνησης ε, μέχρι αυτές που είναι αντίθετες. Έχουν ενισχυθεί οι διμερείς σχέσεις Βραζιλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλούς τρόπους. Είδαμε στις Κάνες η ομάδα G συνεργάζεται με τη Βραζιλία για τη συγκρότηση αυτού του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ε, ενισχύονται οι δεσμοί λοιπόν και το ίδιο ελπίζω να συμβεί και στις σχέσεις με το Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα με την Επιτροπή μας γιατί μπορεί να ανακύψουν παρανοήσεις, ε, ε, προβλήματα και θα πρέπει να δώσουμε μία λύση. Στην περίπτωση Μπατίστη, παραδείγματος χάρη, δεν βασιστήκαμε σε διμερή συμφωνία ανάμεσα στη Βραζιλία και την ε, Ιταλία, οπότε η δράση του Κοινοβουλίου και της Ένωσης περιοριζόταν ακριβώς από αυτό, διότι δεν υπήρχε διμερής ε, συμφωνία. Εγγραφόταν το θέμα γενικότερα στις διμερείς σχέσεις Ιταλίας-Βραζιλίας και ε, στο γενικότερο ένομο πλαίσιο της Βραζιλίας φυσικά δεν αμφισβητώ την ορθότητά του. Ε, επίσης, θα ήθελα να μιλήσω για τις απελάσεις. Ε, υπάρχει ένας ε, πρώην βουλευτής, ε, Πορτογάλος, που έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά του κράτους στη Βραζιλία και δεν ξέρουμε αν θα εκδοθεί ε, διότι υπάρχουν οι συμφωνίες των πορτογαλόφωνων χωρών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ισχύει. Δεν θα ήταν πιο σωστό να υπάρχουν συμφωνίες ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρυθμίζουν την έκδοση των ε, καταζητούμενων. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση ω προ τη μετανάστευση. Όπως είπατε αντιστρέφονται τώρα οι μεταναστευτικέ ε, ροές ε, και αυτό δεν το γνωρίζουν ακόμη οι λαοί των ευρωπαϊκών χωρών ούτε καν όλοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά σίγουρα πηγαίνουν περισσότεροι πλέον Ευρωπαίοι στη Βραζιλία από ότι Βραζιλιάνοι στην Ευρώπη. Επιστρέφουν επίσης ε, Βραζιλιάνοι μετανάστες στη χώρα και ε, σε θελούσια βάση συνεχίζεται η επάνωδος των Βραζιλιάνων που είναι στην, στο Βέλγιο, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, ε, χάρη στη δράση διεθνών οργανώσεων που ε, βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους κατά την θελούσια επάνωδό τους στη χώρα. Λοιπόν, ε, για την Πορτογαλία και την ε, Ισπανία. Ούτως ή άλλως ε, για τη μετανάστευση ε, είναι βασικός προορισμός η Βραζιλία. Δηλαδή οι πτυχιούχοι κυρίω, γιατί πρόκειται για συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις μεταναστεύουν προς τη Βραζιλία, οι αρχιτέκτονες, πιο συγκεκριμένα δημοσιογράφοι, φεύγουν συχνά για να κατασταθούν στη Βραζιλία, υπάρχουν προγράμματα φοιτητικών ανταλλαγών κτλ. Τώρα, λόγω των προβλημάτων, ε, η κοινή γνώμη δεν ασχολείται τόσο πολύ με την αντιστροφή αυτών των μεταναστευτικών ροών, η οποία όμως καθιστά απαραίτητη μια συμφωνία ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία πολύ σύντομα ερωτήματα τώρα. Θα ήθελα να σχολιάσετε διεξοδικότερα τι ε, κοινέ ε, δράσει που θα μπορούσαν ενδεχομένω να αναλάβουν από κοινού η Βραζιλία και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη διαφθορά και την καταπολέμηση τη νομοποίηση ε, του χρήματο από παράνομε δραστηριότητε. Ποιε είναι αυτέ οι νέε δράσει λοιπόν που θα μπορούσαν να ληφθούν από κοινού σε αυτόν τον τόσο σημαντικό τομέα. Επίση, τι πιστεύετε για την καταπολέμηση του σεξουαλικού τουρισμού η Βραζιλία πρέπει ίσως να συμμετάσχει κατά τη γνώμη σας στις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα συμβαίνουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, για τις πτήσεις προς Βραζιλία ε, πρέπει να προστατευτούν τα ατομικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών και πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρον εφόσον ε, ασχολούμαστε τώρα με τα PNR e για τα ε, δεδομένα των επιβατών, δηλαδή στις πτήσεις προς ε, τις ΥΠΑ να αρχίσουμε αντίστοιχες εργασίες και για την Βραζιλία. Θα έπρεπε ε, να έχουμε ρίξει σωστά τα θεμέλια και όχι να ασχολούμε θα με κατακαιρματισμένο τρόπο και να μιλάμε πότε για το SWIFT, πότε για το PNR. Ε, χρειαζόμαστε ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας ατομικών δεδομένων ε, που θα χαρακτηρίζει τις διμερεί σχέσεις ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι κάτι το απαραίτητο για να προστατεύσουμε τα ατομικά δεδομένα και των Ευρωπαίων και των Βραζιλιάνων. Σα ευχαριστούμε. Κυρία Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Νομίζω ότι γνωρίζω τη χώρα σας. Είναι μια χώρα που θαυμάζω. Έχω επισκεφτεί τη χώρα σας πολλές φορές ε, και θεωρώ ότι σε θέματα υποδοχής και διατήρησης της ειρήνης θα μπορούσε να διδάξει πολλά και σε εμά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια ειρηνική χώρα ε, σε σύγκριση δε και με πολλές άλλες χώρες ε, και αυτό διαφαίνεται στη διάρκεια της ιστορίας της. Πρόκειται για μια χώρα που θαυμάζω. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα όσα άκουσα στην παρουσίασή σας για την τρομοκρατία και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ως παγκόσμιο στόχο. Αναφερθήκατε επίσης στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και χαίρομαι ιδιαίτερα που υποστηρίζετε όλες τις συμβάσεις καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα της τρομοκρατίας γιατί είμαι Ισπανίδα και η χώρα μου έχει χτυπηθεί πάμπολες φορές και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα σταματήσει. Ε, να είναι θύμα της τρομοκρατίας. Εδώ και πολλά χρόνια βέβαια ζω στην Ιταλία και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ευαισθησίες των Ιταλών γιατί και αυτοί πλήχθηκαν από την τρομοκρατία όπως γνωρίζετε με τις ερυθρές ταξιαρχίες οι οποίες ε, οδήγησαν σε πολλά δάκρυα και τρομοκράτησαν έναν ολόκληρο λαό. Και ε, υπάρχει και ένα θέμα το οποίο γνωρίζετε και εσείς και το γνωρίζουν ε, και οι άλλοι συνάδελφοι. Ένας εκ των μελών των Ερυθρών Ταξιραρχών ήταν ο Μπατίστη, ο οποίος ε, σκότωσε έναν άνθρωπο με το 14χρονο γιο του και ε, πρόκειται για μια ιστορία την οποία γνωρίζω προσωπικώς. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ε, μείνει ούτε μία μέρα στη φυλακή για τα εγκλήματά του και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έκαναν την έκδοσή του οι βραζιλιανικές αρχές παρά το αίτημα της Ιταλίας. Εγώ ε, στην καλή βούληση των Βραζιλιανών και θα πρέπει να κάνετε μία προσπάθεια να μας εξηγήσετε τα ανεξήγητα, διότι για μας είναι ανεξήγητο. Για μένα ως άνθρωπο που ασχολούμαι με την τρομοκρατία είναι ανεξήγητο. Και θεωρώ ε, ότι είναι δυνα... αδύνατο μία χώρα ειρηνική όπως είναι η Βραζιλία να υποδέχεται έναν τρομοκράτη σαν τον Τσέζαρη Μπατίστη. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όση ώρα θέλετε. Αλλά θα ήθελα να σας πω και επιτρέψτε μου, δεν θέλω να σας προσβάλλω, ότι το να διατηρείτε αυτό τον εγκληματία σημαίνει ότι εγκληματείτε και εσείς. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στην Ιταλία για να πληρώσει για τα εγκλήματα που διέπραξε. Και νομίζω ότι στην περίπτωση του Τσέζαρε Μπατίστη δεν υπήρχε η πολιτική βούληση για να επιληθεί το ζήτημα. Και επειδή εσεί αναφέρεστε σε καταπολέμηση τη τρομοκρατία και καταπολέμηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, των ανθρωπίνων, και διατήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε αυτή την περίπτωση οι πράξει είναι αντίθετε στα λόγια και θα ήθελα να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Χιμένε Εθαρίλ. Τώρα ο Πρέσβη έχει χρόνο για να απαντήσει σε ερωτήσει που ετέθησαν, ιδιαίτερα σε αυτή την υπόθεση η οποία απασχόλησε πολλέ από τι παρεμβάσει, την παρουσία στη Βραζιλία του γνωστού τρομοκράτη Τσέζαρε Μπατίστη, ο οποίο έχει ομολογήσει και τα εγκλήματά του. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Α αρχίσω ευχαριστώντας σας ε, για τις παρεμβάσεις σας. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση που αποτέλεσε αντικείμενο δύο παρεμβάσεων. Κατ' ουσίαν και κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι ένα διμερές ε, ζήτημα ανάμεσα στην Ιταλία και τη Βραζιλία αυτό συγκεκριμένο. Έτσι, ε, το, ε, αυτό θεωρούμε εμείς και συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Μιλάμε εδώ για χώρες, ε, αυτό ισχύει και για την Ιταλία και για την Βραζιλία, που είναι δημοκρατικές. Ε, υπάρχει, υπάρχουν ε, νόμοι, κανονισμοί και το πρώτο που πρέπει να γίνει, σε αυτή την περίπτωση και σε οποιαδήποτε ε, περίπτωση, είναι να τηρήσουμε αυτές τις αποφάσεις, κυριαρχικές αποφάσεις κάθε κράτους και την νομοθεσία που έχει θεσπίσει. Δεν υπάρχει νέα αίτηση έκδοση ε, προς την Ιταλία. Πριν από χρόνια ζήτησε η Βραζιλία από την Ιταλία την έκδοση ε, ενός καταζητούμενου ε, του Σαλβατόρε Κατσόλα, διότι διαβίωνε στην Ιταλία ενώ καταζητεί το από την δική μας δικαιοσύνη. Δεν έγινε η έκδοση, οι Ιταλικές αρχές αποφάσισαν να μην τον εκδώσουν. Τελικά το 2008 συνελήφθη στο Μόνακο, έφυγε από την Ιταλία, πήγε στο Μονακό και επειδή είχε λάβει ένταλμα σύλληψης Ιντερπολ, συνελήφθη και εξεδόθη. Ε, πρόσφατα στον τύπο διάβασα για μία περίπτωση ενός ε, Λατινοαμερικάνου πολίτη που είχε ε, ε, καταδικαστεί τη δεκαετία του 70 για ανθρωποκτονία στη ΣΥΠΑ, ο οποίος συνελήφθη στην Πορτογαλία, αλλά η πορτογαλική δικαιοσύνη απέρριψε την αίτηση έκδοσης διότι βάσει του δημοσιεύματος είχε ήδη αποκτήσει την πορτογαλική εθνικότητα με εντελώς διαφορετικό όνομα όμως. Αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι χαρακτηριστικές γιατί ε, όπως σας είπα στην αρχή πρόκειται για διμερές ζήτημα ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιταλία. Δεν είναι διμερές ζήτημα ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και οι δύο αυτές περιπτώσεις ε, δείχνουν ότι ορισμένες φορές ε, κάποιοι είμαστε στο ένα στρατόπεδο ε, και σε άλλες περιπτώσεις είμαστε στο αντίθετο στρατόπεδο. Αυτό συμβαίνει για, όλες, για όλα τα κράτη δικαίου. Ίσχυε για τη Βραζιλία, την Ιταλία, την Ισπανία, για όλες τις χώρες. Άρα θα πρέπει ξαναλέω να γίνονται σεβαστές οι κυριαρχικές αποφάσεις αυτών των ε, κρατών δικαίου. Δεν πρόκειται να κάνω άλλες παρατηρήσεις. Νομίζω επαρκεί αυτή η τοποθέτηση. Για το θέμα των ε, θεωρήσεων, το οποίο ε, σχολίασε ο αξιότιμος βουλευτής ε, και σχολίασα και εγώ στην πρώτη μου παρέμβαση. Προσθέσατε κι εσείς κάποια στοιχεία ε, λοιπόν, σχολίασα στην ε, παρέμβασή μου τους λόγους για τους οποίους διαπραγματευτήκαμε μια συμφωνία και εσείς ε, δώσατε κάποια άλλα στοιχεία. Η πρώτη εναλλακτική λύση, όταν Αρχίσαμε να εξετάζουμε το θέμα της ε, μη εφαρμογής ε, από πλευράς αυτών των τεσσάρων χωρών ε, των διατάξεων περί απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Μας έγινε γνωστό τέλος πάντων από συγκεκριμένους βραζιλιάνους πολίτες και για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση υπογράφουμε αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Εγώ όταν έφτασα το 2008 ήρθα σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσώπους αυτών των τεσσάρων χωρών για να διαπραγματευτούμε διμερεί νομικά μέσα ακριβώς όπως αυτά που είχαμε με τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, νωρίτερα. Η απάντηση που πήρε είναι ότι υπάρχουν ε, διάφορες αλλαγές ε, ως προς τη διαδικασία ενσωμάτωσης των αλλοδαπών και ότι είναι θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών και ότι συντονίζει τη δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι υπάρχει μια συμφωνία που ισχύει για όλες τις χώρες εκτός ε, από δύο. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε μία συμφωνία ε, που θα λαμβάνει υπόψη τις πρώτερες διμερείς συμφωνίες για την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης Οι συμφωνίες αυτές ε, θα πρέπει να ισχύουν για διαμονή τρίμηνη με δυνατότητα παράτασης ε, τρίμηνης επίσης. Η όλη διαδικασία ήταν εξαιρετικά αργή καθότι περίπλοκη και στην ε, περίπτωσή μας εξάλλου ομολογώ ότι ήταν η πρώτη φορά που χρειάστηκε να εκπονήσουμε και να προσπογράψουμε μια τέτοια συμφωνία με ένα ευρύτατο φάσμα χωρών, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πέρυσι, και ως προς την υπογραφή των ε, συμφωνιών με τις υπόλοιπες τέσσερις χώρες ε, που προανέφερα και εν ώψη της ε, Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βραζιλίας είχαμε εξετάσει το ενδεχόμενο να προσυπογράψουμε τη συμφωνία. Υπήρξαν όμως τεχνικά προβλήματα, μετάφραση, διάφορα διαδικαστικά ζητήματα και τελικά δεν υπεγράφει αυτή η συμφωνία. Επίσης είχαμε εκείνη την περίοδο ε, προεκλογική εκστρατεία στην ε, Βραζιλία, καθυστέρηση η διαδικασία, σημειώθηκε και άλλη καθυστέρηση γιατί σας είπα ότι εξετάζονται αυτή η συμφωνία για τις τέσσερις χώρες από την ε, γερουσία μας. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ήδη έχει τεθεί σε ισχύ η άλλη συμφωνία που δεν χρειάζεται κύρωση από τη Γερουσία. Πρόκειται, όπω σα έλεγα προηγουμένω, για τη συμφωνία για τα διπλωματικά ε, επίσημα και υπηρεσιακά ε, διαβατήρια. Ξέρετε, είναι σαφώ διαχωρισμένη η εκτελεστική από την νομοθετική εξουσία στη Βραζιλία και άρα δεν μπορώ εγώ να προδικάσω πότε ακριβώ θα ολοκληρωθεί η εξέταση αυτή τη συμφωνία από το, τη Γερουσία μα. Ξέρουμε όμως ότι ε, το γοργόν και χάριν έχει, διότι έτσι θα μπορέσει να τεθεί ταχύτατα σε εφαρμογή ε, η συμφωνία και ούτως ή άλλως καταβάλουμε άοκνες προσπάθειες για να το επιτύχουμε, για να ρυθμίσουμε αυτή την κατάσταση το ταχύτερο δυνατόν. Τώρα σε σχέση με αυτά που μας είπε ο βουλευτής Ρούι Βάρης, σχετικά με την, ε, ε, το ενδεχόμενο υπογραφής νέων συμφωνιών ε, σε διάφορους τομείς που αναφέρατε. Αναφέρθηκατε συγκεκριμένα στη μετανάστευση, μιλήσατε για το σεξουαλικό τουρισμό, για την καταπολέμηση διαφθοράς, για την καταπολέμηση νομοποίησης, χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Μιλήσατε για ε, ε, συμφωνίες αυτού αυτούς τους Ναι, αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να εξεταστεί από αμφότερες πλευρές. Ε, αυτή τη στιγμή δεν έχω καμία εντολή για να συζητήσω μαζί σας για αυτές τις συμφωνίες. Πιστεύω ότι το εκτελεστικό σκέλος της εξουσίας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν υπήρξε δηλαδή καμία αίτηση, να σας το πω αλλιώς, προς τη Βραζιλία για συγκεκριμένες συμφωνίες στους τομείς αυτούς ε, ε, για τις μεταναστευτικές ροές, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να λύνουμε τα προβλήματα όταν αυτά ανακύπτουν. Ναι. Υπήρξαν ε, διάφορα προβλήματα όταν παραδείγματο χάρη πήγανε Βραζιλιάνοι στην ε, Πορτογαλία στις αρχές δεκαετίας 80 ή και 90 και θυμάμαι συγκεκριμένες περιπτώσεις οδοντιάτρων Βραζιλιάνων που δυσκολεύονταν ε, στη διαμονή τους και στην εργασία τους στην Πορτογαλία λόγω των ε, απαιτήσεων ακαδημαϊκής ε, κατάρτισης που απαιτείται και είναι πάρα πολύ περίεργο ξέρετε γιατί στη Βραζιλία ε, ήδη με το που μπαίνουν στην οδοντιατρική οι φοιτητές αρχίζουν εξ αρχής και τα μαθήματα για να γίνουν οδοντίατροι. Αρχίζουν με ενώ στην Πορτογαλία πρώτα γίνονται ιατροί και μετά οδοντίατροι. Και εκεί έξω και το πρόβλημα της αναγνώριση των πτυχίων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Ξέρετε πόσο παλιέ είναι οι σχέσει ανάμεσα στι δύο χώρε και είμαι πεπισμένο θα βρούμε λύση για αυτά τα προβλήματα. Σήμερα έχουμε το αντίστροφο πρόβλημα, δηλαδή ε, Πορτογάλοι που θέλουν να έρθουν να εργαστούν στη Βραζιλία, αλλά έχουν ε, κάνει τη φοιτησή του σε πορτογαλικά ε, ακαδημαϊκά ιδρύματα και δεν είναι αναγνωρίζονται τα πτυχία τους. Ελπίζουμε να βρούμε μια ικανοποιητική λύση για να ρυθμίσουμε τα προβλήματα ε, ε, και όλα τα προβλήματα ε, όταν ανακύπτουν, όπως σας είπα για τις νέες δράσεις, για το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών, νομίζω θα πρέπει να εξετάσουμε με μονομένες ε, περιπτώσεις. Δεν νομίζω ότι τώρα μπορώ να αποφανθώ για συγκεκριμένα ζητήματα, διότι δεν υπάρχουν διαβουλεύσεις ε, προς το παρόν για την ε, προετοιμασία και την ε, επικύρωση τέτοιων ε, συμφωνιών. Είναι μάλλον υποθετικό το ερώτημά σας και δεν μπορώ να τοποθετηθώ περαιτέρω καθότι πρόκειται για ένα υποθετικό σενάριο. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη για την παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή μας κατόπιν προσκλήσεων των μελών. Ε, και σας ευχαριστούμε και για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Ο κύριος Γιακολίνο θέλει να πει κάτι ακόμα. Πολύ σύντομα, για τις ε, τουριστικές θεωρήσεις, ε, κύριε Πρέσβη, δεν μας απαντήσατε. Υπάρχει διάκριση μεταξύ πολιτών κάποιων κρατών μελών σε σχέση με κάποιους άλλους, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κύρωση. Για την περίπτωση Μπατίστη δεν το συζητάω άλλο. Εκτός μικροφώνου, απαντά ο Πρέσβης. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη, άκουσα απευθεία στα Ιταλικά γιατί σπούδασα εγώ Ιταλικά πολλά χρόνια και προσπαθώ να σας καταλάβω, προσπαθώ να ακούω και να σας καταλάβω στη μητρική σας, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι σας κατάλαβα ακριβώς. Θα ρωτήσω εδώ το συνεργάτη μου. Ένα λεπτό. Επαναλαμβάνω πολύ σύντομα. Από τον Ιούνιο του 2011 οι θεωρήσεις διαβατηρίων για τουριστικούς σκοπούς, ε, για ε, προσωπικούς λόγους, έχουν περιοριστεί στις 90 μέρες για τους Ιταλούς πολίτες. Θα έπρεπε να το έχω πει ήδη. Η σχέση ανάμεσα στην Ιταλία και την Βραζιλία είναι ε, εξαιρετικά ευρεία, εξαιρετικά παλιά. Ε, πάνω από 30.000 ε, ε, άνθρωποι ε, μπορούν να αποκτήσουν την Ιταλική υπηκότητα. Βλέπετε ότι υπάρχουν στενές σχέσεις, υπάρχουν συγγενείς, παιδιά, νύψια Υπάρχουν στενές οικογενειακές σχέσεις ανάμεσα σε διάφορες κοινότητες των χωρών μας. Και για τις θεωρήσεις σύντομης διάρκειας, στα πλαίσια της συμφωνίας που έχουμε με την Ιταλία και μην ξεχνάτε ότι θα εφαρμοστούν και αυτές οι δύο νέες συμφωνίες στις οποίες αναφερθήκαμε νωρίτερα. Προβλέπεται λοιπόν ότι ε, η διαμονή 90 ημερών είναι κατοχυρωμένη με πιθανότητα παράταση σε κάτω 90 ημέρες. Ε, και αυτό ισχύει για όλους ε, τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτές τις δύο συμφωνίες που υπογράψαμε πέρυσι, αυτό προβλέπεται ακριβώς. Από πλευράς της Βραζιλίας μπορεί να προβλεφθεί ε, παράταση ε, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με τις διατάξεις για τις επιστροφές μετά τις υποχρεωτικές επτήσεις. Δεν ξέρω τι ισχύει σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά σίγουρο είναι ότι υπάρχει πιθανότητα παράτασης κατά 90 ημέρες. Δηλαδή, εάν ένας Βραζιλιάνος θέλει να μείνει στην Ευρώπη, αντίστοιχα ένας Ευρωπαίος ε, να μείνει στη Βραζιλία για πάνω από τρει μήνες, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. πλαισιώνεται αυτή η περίπτωση από άλλε συμφωνίε. Κάποιο που θέλει να πάει να δουλέψει σε μια άλλη χώρα. Ε, και άρα ε, ο στόχος δεν είναι τουρισμός, ε, είναι οικονομικός μετανάστης. Αν θέλει κάποιος λοιπόν να παραμείνει και ε, στη χώρα διότι άλλαξε γνώμη και θέλει να εργαστεί θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση και να τεκμηριώσει την αίτησή του ε, για μία περίοδο που υπερβαίνει αυτές τις 90 συν 90 ημέρες. Ε, ε ο κ. Γιακολίνο με την απάντηση. Τα νέα που έχουμε εμείς ίσως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα διότι από 1η Ιουλίου σε όλες τις θεωρήσεις που αφορούν τους Ιταλούς υπάρχει μια σφραγίδα που λέει χωρίς παράταση. Δηλαδή οι 90 αυτές οι μέρες είναι χωρίς παράταση. Ε, Ας ελπίσουμε αυτά τα οποία διαβάσαμε σε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα στα τέλη του Σεπτεμβρίου ε, να έχουν επιληθεί και να ισχύουν αυτά τα οποία μας είπε ο πρέσβης. Δηλαδή να είναι 90 συν 90 μέρες και να είναι δυνατό αυτό το ενδεχόμενο. Κάτι τελευταίο πολύ σύντομα. Ευχαριστώ τον πρέσβη. Κοιτάξτε να δείτε κύριε Πρέσβη, εμείς μαζί με τον κύριο Μπουσουτήλ και άλλους συναδέλφους πήγαμε με μια αντιπροσωπεία στη Σικελία και επισκεφθήκαμε διάφορα κέντρα προσφύγων. Και με τα άτομα που συναντήσαμε, τα όσα παρακολουθήσαμε, ιστορίες που ακούσαμε των προσφύγων, ε, είναι πολύ διαφορετικά από την υπόθεση Μπατίστη, την οποία εσείς ε, ε, αντιλαμβάνεστε ως έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς έχει ζητήσει καταφύγιο στη χώρα, ενώ είναι ένας εγκληματίας ο οποίος θα έπρεπε να εκδοθεί και να μπορέσουν να τηρηθούν αυτές οι διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των χωρών και ελπίζουμε να βρεθεί μια λογική και σωστή λύση. Κύριε Πρέσβη, μια τελευταία κουβέντα. Είπα ότι έπρεπε να πω.